Shall we start? Ladies and gentlemen, please stay. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σας, ξανακαλωσορίζω. Είναι η κυρία Λουέγκα και ο κύριος Μωράς που δεν μπορούν να είναι σήμερα εδώ γιατί έχουν ε, υποχρεώσεις ε, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας στη Βιέννη. Έχουμε τον εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Μικρή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και πρώην εισηγητή της ε, Europol που θα, θα τους αντικαταστήσει. Καλημέρα κύριε είστε μέρα. Εύχομαι να έχουμε μια καλή συνεδρίαση. Το όνομα μου είναι Κρίστιαν Μπούχμαν. Είμαι ο πρόεδρος της ε, ε, του Κοινοβουλίου της Αυστρίας, του Συμβουλίου της Αυστρίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και ήμουνα και περιφερειακός υπουργό. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας δείξω. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από Σουηδικά και επίσης να σας πω στις ε, διαβουλεύσεις της Τρόικα είχαμε αποφάσεις για τις οποίες θέλω να σας ενημερώσω συνάδελφοι. Θέλω να σας πω ότι η Προεδρική Τρόικα ενέκρινε το, το καταστατικό με πλήρη την κτήμα ελέγχου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού της Europol και μέχρι την επόμενη συνεδρίαση στη 15 Φεβρουαρίου του 2019 οι συνεδριάσεις της ε, Europol είναι παρατηρήσεις που δεν ψηφίζει Τα ευρήματα θα σας ε, παραδοθούν γραπτός. Προτείνανε τον κύριο Σμετάνοφ για αυτή την πολύ σημαντική λειτουργία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος από εσάς έχει αντίθετη γνώμη με αυτή την πρόταση. Δεν βλέπω, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο κύριος Βεντάτοφ είναι εκπρόσωπός μας, λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφοι, θα περάσουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη και θα ξεκινήσουμε με μία ανταλλαγή απόψεων με τον ε, επόπτη Προστασία δεδομένων. Προτού δώσω το λόγο, πρωτού μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση, θα σας πω πώς ε, θα είναι η συνεδρίαση σήμερα. Θα έχουμε το ίδιο μοντέλο με χθες, πρώτο με χθες. Θα έχουμε δύο από τις εθνικές ε, αντιπροσωπείες ε, και δύο από το Ευρωκοινοβούλιο μέχρι να εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τις καρτέλες να τις παραδώσετε στο Προεδρείο. Να σας πω επίσης ότι τόσο οι εκπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίου όσο και του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να συμπληρώσουν τις καρτέλες όταν θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Δύο λεπτά χρόνος ομιλίας. Θα ήθελα να περιστείτε σε αυτόν. Μπορεί να προσαρμόσουμε τον χρόνο ανάλογα με το πόσο χρόνο θα μας περισσέψει για να μπορέσουν όλοι να πάρουν τον λόγο. Ο κύριος Βιερόφσκι, Ευρωπαϊκός Υπόπτης Προστασίας Δεδομένων, ο λόγος εσάς, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτήν την συνάντηση και να σας ενημερώσω όσον αφορά τις εποπτικές αρμοδιότητες που έχουμε απέναντι στην Europol. Όπως γνωρίζετε, ο επόπτης είναι επόπτης όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς σε σχέση με την προστασία. Και συγχρόνως, 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν 28 διαφορετικές δικαιοδοσίες σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, διότι η νομοθεσία όσον αφορά την εποπτεία του τι γίνεται δηλαδή με την τήρηση της νομοθεσίας είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την άλλη μεριά όμως πάρα πολλές αρμοδιότητες είναι των εθνικών αρχών. Οπότε η εποπτεία, ο έλεγχος δηλαδή όλων των αρχών ε, και των ε, αρχών έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία μας στέλνουν οι υπηρεσίες αυτές, στην Europol δηλαδή. Από το 2017 που πτεύουμε πλήρως στην Europol όσον αφορά τα δεδομένα, κάτι το οποίο μας έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερα καρποφόρα συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο διαχείρισης, σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή με εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με το έργο της Europol επιτόπου. Είχαμε μια επιχειρησιακή επίσκεψη ήδη το 2017, έκτοτε όμως ξεκίνησε στην πράξη το έργο μας. Με δύο επιθεωρήσεις που κάναμε, η μία ολοκληρώθηκε μετά την τελευταία συνάντηση της ομάδας σας και η δεύτερη ε, επιχείρησή μας ολοκληρώθηκε τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε συναντήσεις με τη Europol που οργανώνονται ε, κάθε δεύτερο μήνα και η τελευταία έγινε χτες, χτες, εδώ στις Βρυξέλλες. Εμείς ε, έτσι είμαστε σε επαφή με την ε, Europol και το προσωπικό μας ε, εποπτείας έχει έτσι δυνατότητα να συζητά διάφορα καυτά ζητήματα αλλά και νέα σχέδια με τους αξιωματούχους της Europol αλλά και πιο συγκεκριμένα της μονάδας που ασχολείται με την προστασία δεδομένων. Επίσης έχουμε αναπτύξει και καρποφόρα συνεργασία με την Europol σε υψηλό επίπεδο. Και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί με τον εκτελεστικό διευθυντή της Europol τον Ιούλιο. Τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία γίνονται τώρα είναι, όπως είπα, επιθεωρήσεις και συνεργασία στην πράξη. Η πρώτη επιθεώρηση έγινε το Δεκέμβριο του 2017 και το πεδίο εφαρμογή ήταν να γίνει έλεγχος νομικός, διοικητικός. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι ελέγχουμε στου στους ελέγχους αυτούς, στις επιθεωρήσεις αυτές, ε, τις δραστηριότητες του προσωπικού. Το πιο σημαντικό όμως όσον αφορά το έργο της Europol είναι η τεχνική και νομική ανάλυση που κάνουμε επιτόπου. Από νομική άποψη πρόκειται για τα δεδομένα, την επεξεργασία τους σε δύο επιχειρησιακές ε, αναλύσεις για μετανάστες, για διακίνηση ηρωίνης κλπ. Η τεχνική πτυχή τώρα, τεχνική έλεγχη έχουν να κάνουν με τον έλεγχο της ε, προστασίας των πληροφοριών και των ε, κανόνων και των πρακτικών λύσεων που συνδέονται με την διατήρηση δεδομένων. Η έκθεση στάλει στη Europol το Μάιο με 45 συστάσεις. Οι περισσότερες από αυτές ήταν ε, τεχνικού χαρακτήρα, πρόκειτο για διορθώσεις ή για ε, συστάσεις που κάναμε, προτάσεις. Δεν βρήκαμε κάτι το οποίο θα μας υποχρέωνε να μπούμε στη διαδικασία μιας επίσημης διερεύνησης όπως θα μπορούσε να κάνει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Οι συστάσεις μας αυτές, λοιπόν, ελέγχονται από τον ε, Ευρωπαίο Επόπτη για την προστασία των δεδομένων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτή ήταν η πρώτη μας ε, επιθεώρηση. Η δεύτερη συνδεόταν με τα συστήματα ΣΥΣ, πληροφοριών δηλαδή, όσον αφορά ανήλικες και είχε να κάνει και με ελέγχους όσον αφορά μετανάστες στα hot spots. Και αναλύσαμε επίσης και στοιχεία για ταξιδιώτες. Τεχνικά μιλώντας ε, λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε το θέμα της διαχείρισης, της ασφάλειας δηλαδή στην διαχείριση των δεδομένων. Τα διοικητικά ε, στοιχεία και οι έλεγχοι έγιναν βάσει επιλογής. Η Europol έχει ήδη εγκρίνει τα πρακτικά της επιθεώρησης αυτής και συντάσσεται σχετική έκθεση και συστάσεις. Το επόμενο βήμα για μας είναι η επιθεώρηση που σχεδιάζομαι για τα τέλη του 2018, που θα επικεντρωθεί στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η Europol παίζει και εδώ ένα σημαντικό ρόλο. Τώρα το άλλο σκέλος του έργου του Ευρωπαίου Πόπτη Προστασίας Δεδομένων που έχει να κάνει με την επιθεώρηση της Europol είναι η οργάνωση της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές, με τους εθνικούς επόπτες προστασίας δεδομένων δηλαδή. Εδώ οι εργασίες γίνονται σε ομάδες συνεργασίας. Υπάρχει ένα συμβούλιο που συμμετέχει ο επόπτης προσωπικών δεδομένων, Ευρωπαίος δηλαδή, και 28 εθνικές αρχές από τις 28 χώρες. Εκδώσαμε και γνωμοδοτήσεις για διάφορα προγράμματα και για διάφορες νομικές πράξεις που προετοιμάζονται ε, τώρα. Θα το ξέρετε και το συζητήσαμε και στη Σόφια. Έχουμε γνωμοδότηση για τη συνεργασία με ξένους εταίρους, τους Europol δηλαδή, με ξένους εταίρους, που σημαίνει κυρίως διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν με την Αλγερία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τουρκία για δεχομένω ανταλλαγή δεδομένων με τις χώρες αυτές. Αποτέλεσε και αυτό μέρος των συζητήσεών μας στη Σόφια. Ξέρετε ότι διαπραγματευόμαστε εντολή που ενέκρινε το Συμβούλιο που συμπεριλαμβάνει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη για την προστασία των δεδομένων κυρίως όσον αφορά τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών στις διάφορες χώρες, αλλά και την υποχρέωση επέκταση των περιορισμών όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων με αυτές τις χώρες. Όπως επίσης και το θέμα της άρσης των συμφωνιών αυτών για τα δεδομένα. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υπάρχουν γνωμοδοτήσεις από την πλευρά μας, μεταξύ άλλων για τη συνεργασία της Europol μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα η συνεργασία με την Frontex, Είχαμε διαβούλευση όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Europol και Frontex. Το Σεπτέμβριο έγινε αυτό που μας πέρασε. Επίσης, είχαμε διαβουλεύσεις και για τον ρόλο της Europol στην επεξεργασία δεδομένων και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο ασχοληθήκαμε με την συνεργασία όσον αφορά τις ε, πληροφορίες για τα οικονομικά δεδομένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία. Υπάρχει συντονιστικό συμβούλιο στη Europol για αυτά. Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι και για νομικά θέματα και σε υψηλό επίπεδο υπάρχει συνεργασία και κυρίως πρακτικά. Η συνεργασία μας με το Europol πηγαίνει σε βάθος, πηγαίνει πολύ καλά. Παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Ε, βλέπουμε ότι αντιδράει η Europol κάθε φορά που εμείς εκφράζουμε κάποιες αφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα τα συστήματα πληροφοριών. Ε, συμβαίνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ζητάμε περισσότερες πληροφορίες, αφισβητούμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πάντω ότι οι απαντήσεις που έχουμε από τη Europol είναι πάντα πολύ καλές, ικανοποιητικές και πάντα βρίσκουμε λύσει ακόμα και αν μερικέ φορές ε, χρειάζονται επιπλέον επενδύσει από τη Europol. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και την ορθή διαχείριση του χρόνου, κύριε Ντιέ Ντεμέρα. Θα προεδρεύσει τη συνεδρία σα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τον ε, κύριο Βιβυρόφσκι για την παρουσίασή του όσον αφορά την προστασία δεδομένων από πλευρά της Europol. Θα δώσουμε τώρα το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Γκρούλιτς από την Τσεχία. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι η τσεχική δημοκρατία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη φιλοδοξία, συγκεκριμένη φιλοδοξία όσον αφορά τις εργασίες αυτής της ομάδας Όμως είναι παράξενο το ότι δεν μπορούμε να εκλέξουμε έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Europol. Τρία χρόνια έχουν περάσει, τρία χρόνια ετοιμάσαμε το, χρειαστήκαμε για να ετοιμάσουμε τον εσωτερικό κανονισμό. Και δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε το θέμα. Και αυτό είναι πολύ πολύ παράξενο. Ο κύριος Γρουλίτς. Πρέπει να πω ότι η μερίσια διάταξη στο σημείο αυτό προβλέπει την ε, συζήτηση όσον αφορά την παρουσίαση που μόλις ακούσαμε του κύριου Βιβυρόφσκι για την προστασία δεδομένων από πλευρά της Europol. Αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε έχει δύο-τρία διαφορετικά σενάρια στα πλαίσια της Τρόικα. Στην αρχή ο πρόεδρος Μπούκμαν αναφέρθηκε στο σημείο αυτό. Προτείνω με κάθε συμπάθεια να διαβάσετε το άρθρο 14, σημείο 4 του κανονισμού και εκεί θα βρείτε απάντηση στις αμφιβολίες σας και στις ερωτήσεις σας. Τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Χετίνος από την Κύπρο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Καλημέρα σας. Με αφορμή το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο Ιούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων συνομιλιών σχετικά με ανταλλαγέ προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Europol με τρίτες χώρες, συγκεκριμένα η Ορδανία, Τουρκία, Ισραήλ, την Ισία, Μαρόκο, Λίβανο, Αίγυπτο και Αλγερία, που στόχο έχουν την αποτροπή και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, στο οποίο υπογραμμίζεται η ανάγκη για μια εκτίμηση αντικτύπου σε βάθος όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι εν λόγω ανταλλαγές δεδομένων, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε εάν τελικά η Κομισιόν, εάν γνωρίζετε, αν έχετε εσείς την πληροφορία, θα προβεί, έχει την πρόθεση να προβεί σε τέτοια ανάλυση αντικτύπου. Και με την ευκαιρία να επαναλάβω την ανησυχία την οποία εξέφρασε χθε ο συνάδελφός μου ο κύριος Δημητρίου σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τις ισχυρές επιφυλάξεις που διατηρούμε για τη συμπερίληψη της Τουρκίας στις μεσογειακές χώρες με τις οποίες, ε, με ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία ανταλλαγή προσωπικών ε, δεδομένων. Επαναλαμβάνουμε το γεγονό ότι η χώρα αυτή διατηρεί χαμηλό επίπεδο προστασία δεδομένων και ότι η Τουρκία δεν συνεργάζεται με την Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κετινό. Μετά ο κύριος Βιδιορόφσκι θα απαντήσει δίχως άλλο. Η κυρία Καραμάλ τώρα έχει το λόγο από την Γαλλία παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι απλή ερώτησή μου και αφορά τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τρίτες χώρες για συμφωνία που αφορά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ των χωρών αυτών και της Europol. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε και υποβάλλουμε σχετικά την ερώτηση. Εξηγήστε μας τι εγγύησεις έχουμε, τι προβλέπετε, ούτως ώστε τρίτες χώρε να χρησιμοποιούν σωστά τα προσωπικά δεδομένα και να μην διαβάζουν τα στοιχεία σε τρίτε χώρε που δεν είναι εγκεκριμένε να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία. Ποιε αρχέ είναι επιφορτισμένε για την επαλήθευση τη σωστή χρήση αυτών των δεδομένων και διερωτώμεθα επί του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη που είναι κάτοχοι των πληροφοριών και που διαβιβάζουν πληροφορίε στη Europol αν μπορούν να αντιταχθούν, ούτω ώστε κάποιε πληροφορίε να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτε χώρε, διότι θεωρούν ότι αυτέ οι χώρε δεν παρέχουν τα αναγκαία χέγγια για το σεβασμό του κράτου δικαίου. Και τέλο, πιο γενικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν πηγαίνει πολύ μακριά στη φροντίδα που δείχνει για την ασφάλεια, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αστυνομική συνεργασία με χώρες που δεν συμμερίζονται ε, που δενεί ε, τις δημοκρατικές μας αξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Να αντιδράσει ο κύριος Βιβυρόφσκι, να απαντήσει δηλαδή στις τρεις παρεμβάσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όλες μαζί να τις καλύψω, διότι είναι παρόμοιες οι απαντήσεις. Καταρχάς, να τονίσω ότι ο υποπτικό φορέα για τα προσωπικά δεδομένα είναι ο λεκτικό φορέα τη Ευρωπαϊκή Ενώσης Δεν αντιπροσωπεύουμε ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε ξεχωριστό φορέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, εποπτεύουμε τα τεκτενόμενα εκεί. Η άποψή μα για το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια άποψη που αφορά ε, α, α, άλλα θεσμικά όργανα, όχι το δικό μα φορέα. Να πω ότι είδαμε. Ε, πολλούς περιορισμούς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, υπάρχει μια ανάγκη διαφορετική συνεργασίας με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι όπως γνωρίζετε και όπως τονίσαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις άλλωστε, δεν αφορά την αποστολή των, Ευρω... των δεδομένων περί Ευρωπαίων προς τα έξω, αλλά εξετάζουμε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει στοιχεία από τις χώρες με τις οποίες θα συνεργαζόμαστε. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και το ETPS και η ίδια η Europol γνωρίζουν ότι η κατάσταση στις 8 χώρες αυτές διαφέρει εντελώς από τη μια χώρα στην άλλη και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ακολουθήσουμε μία και μοναδική λύση αντιμετωπίζοντας αυτές τις χώρες και ανάλυση των όσων συμβαίνει, συμβαίνουν εκεί και πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα σε κάθε χώρα πρέπει να είναι μια ανάλυση πάρα πολύ ακριβής. Πώς μπορούμε αυτή να εξασφαλίσουμε τη χρήση των δεδομένων στις άλλες χώρες. Ποια είναι τα όρια που ενδεχομένως μπορούμε να επιβάλλουμε για την επεξεργασία των δεδομένων. Ε, βέβαια μπορούμε να εμπιστευθούμε τους ξένους εταίρους, αλλά ακόμα και αν τους εμπιστευόμαστε θα πρέπει να έχουμε την επίσημη συμφωνία και επίσημες λύσεις που θα προβλέπονται στη συμφωνία που θα συναυθεί με την τρίτη χώρα. Ταυτόχρονα, ό,τι και αν αναφέρεται επί χάρτου θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Και αυτό είναι το δυσχερέστερο τμήμα των προσπαθειών και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τον Ευρωπαϊκό ε, Φορέα Εποπτείας των Δεδομένων γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση αυτής της χώρας. Βλέποντας τον κατάλογο των χωρών, να σας πω ότι υπάρχει μια χώρα που έχει σύστημα ασφαλείας δεδομένων ότι είναι χώρες που ελέγχουν την επεξεργασία των δεδομένων μεταξύ τους. Υπάρχουν χώρες όπως το Ισραήλ, υπάρχει αυτή η κατηγορία χώρων. Άλλες χώρες είναι αρκετά καινοφανείς στο σύστημα αλλά έχουν τουλάχιστον μια αρχή προστασία δεδομένων, όπω είναι το Μαρόκο. Μετά έχουμε τι χώρε που απλώ τώρα ξεκινάνε, όπω η Τουρκία και η Τινησία, και χώρε όπου δεν υπάρχει αρχή προστασία δεδομένων για την ώρα, όπω είναι ο Λίβανο, η Ορδανία, η Αίγυπτος και η Αλγερία. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Αν συγκρίνουμε τις υφιστάμενες νομοθεσίες, πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία έχει πολύ νέο καθεστώς υποστασία των δεδομένων που εδράζεται επί πολύ παλαιών παραδειγμάτων από άλλα τμήματα της Ευρώπης. Μοιάζει περισσότερο με τα συστήματα που είχαμε στην Ευρώπη προ 20 αιτίας. Και παρακαλώ επιτρέψτε μου να μην αξιολογήσω ίδιο την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή και τη δυνατότητα να εφαρμοστούν οι νομικές πράξεις ε, που εφαρμόζονται, προβλέπονται στη χώρα. Τι βλέπουμε και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επίτροπης και από πλευράς Συμβουλίου βλέπουμε πολύ ε, ευαίσθητη προσέγγιση όσον αφορά τις συμφωνίες που απαιτούνται από της Ευρωπαϊκής Ενώσης και από την ίδια την Europol. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές αμφιβολίες όσον αφορά την πρακτική χρήση των λύσεων που δημιουργούνται και σε ευρωπαϊκό εποπτικός επόπτης χρήσεως δεδομένων θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο η αδίποτε ανάλυση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την ίδια την Ευρωπόλ γίνεται σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο σε έναν σπουδαίο εμπειρογνώμονα, τον ε, Νικολά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την ΟΕΔΙΟ του 2001 που ανανεώθηκε και και αυτό αυτές οι ε, διατάξεις και για την Europol και για την Eurojust, αλλά αυτό το πλαίσιο δεν ήταν αρκετό για να καλύψουμε και να δώσουμε την απαραίτητη ελευθερία στις διοκτικές αρχές. Η διάδοση των δεδομένων κατά την άποψή μου θα πρέπει να πλησιθεί από πρότυπα χωρίς να περιορίσει περαιτέρω την ελευθερία της Europol. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα θεμέλιο, πλέον μια βάση με την οποία μπορούμε να εργαστούμε ορθά. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε μόνο αν θα πρέπει να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τα δεδομένα όσον αφορά ε, το έργο των ιδιωτικών αρχών και γι' αυτό θεωρώ ότι πλέον έχουμε τη βάση και για τη Europol ώστε να γνωρίζει πότε και σε ποιον μπορεί να μεταδίδει τα δεδομένα και πώς θα τα επεξεργάζεται. Και υπάρχει και ο διαχωρισμός ανάμεσα στο διοικητικό κομμάτι και το οργανωτικό κομμάτι ή το κομμάτι της δίωξης. οι οποίοι ε, ουσιαστικά γνωρίζουν πώς ε, θα ενεργοποιηθούν ανάλογα με τη δικαιοδοσία τους. Αυτό λοιπόν που έχουμε σαν βάση είναι αρκετό θεωρώ για την Europol ε, η οποία ε, ουσιαστικά εμπλέκεται στο κομμάτι της προστασίας δεδομένων και έτσι μπορεί να γνωρίζει τι πρέπει να πράξει. Και της ασκείται έλεγχος. Το θέμα λοιπόν αυτό μπορούμε να το κλείσουμε, να το ολοκληρώσουμε και να αφήσουμε τις αρχές της Europol στην ησυχία τους για να κάνουν τη δουλειά τους εφόσον ήδη έχουν μια βάση πάνω στην οποία μπορούν να εργαστούν. Ευχαριστούμε πολύ, Άξελ. Από το Εθνικό Κοινοβούλιο ακούσαμε τρεις παρεμβάσεις τώρα. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Κινίτσι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, διότι έφτασα δυστυχώς ε, αργά. Είχαμε κάποιες εργασίες σε άλλη συνεδρίαση, όπου εκεί συζητήθηκε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και περίπλοκο της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής και ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι νέα πρόκληση ε, και για το DPS και όχι μόνο για την συμμετοχή, την ανταλλαγή ε, δεδομένων με διάφορους φορείς και ότι χρειάζεται συντονισμό συστημάτων που δεν είναι συντονισμένα και όμορφα και πόροι που δεν είναι συντονισμένοι, αλλά και λόγω περιπλοκότητας ε, διαδικασιών εποπτείας. Έχω μια ερώτηση που σας απευθύνω. Δηλαδή με ποιο τρόπο το, ο, επόπτη, ο επόπτης χρήσεως στοιχείων θα ελέγξει τις εξελίξεις, κυρίως στα πλαίσια της συνεργασίας της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Τι αντίκτυπο μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να έχει αυτή η εξέλιξη και όσον αφορά τη λειτουργία διακοινοβουλευτικού ελέγχου της Europol, μιλώντας για τη λειτουργικότητα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αξιολογούμε και τον αντίκτυπο που θα έχει ο νέο μηχανισμός αυτός. Λοιπόν, σα ευχαριστώ και των προτέρων για την απάντησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Η κυρία Μιτάχ, Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Μια πληρωματική ερώτηση για τον επόπτη προστασία δεδομένων. Είπατε ότι βρίσκεται στη φάση των διαβουλεύσεων και άκουσα από κατάλαβα ότι υπάρχουν ε, προβλήματα στην ανταλλαγή δεδομένων και ότι θα πρέπει να επεκταθεί η Frontex για να μπορεί να έχει διαθέτηση περισσότερο όγκο δεδομένων και η Europol θα πρέπει να μπορέσει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα. Αν δεν λέει χώρα αυτή ότι ε, η ανταλλαγή δεδομένων, δεν θα λάβει μάλλον χώρα αυτή η ανταλλαγή δεδομένων, θα μπορούσαμε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες προς το σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν σε αυτές τις ε, διαβουλευσει. Una pregunta... Πολύ σωστή ερώτηση και πολύ ενδιαφέρουσα. Ο κύριος Παρβιάνεν, Φιλανδία. Παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στη συζήτηση για την ποιότητα αυτής. Η οδηγία περί προστασίας δεδομένων εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος μέλος. Όταν αναφερόμαστε στην προστασία των δεδομένων, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η κατάσταση στα κράτη-μέλη διαφέρει. Όπως είπε και ο πληρωτής επόπτης για τα δεδομένα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι παρόμοιες προδιαγραφές, παρόμοια πρότυπα σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε ένα βαθμό σύγκλησης. Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει συντονισμός βελτίστων πρακτικών στα κράτη-μέλη σε επίπεδο ευρωπαϊκό, διότι η κατάσταση ποικίλει πολύ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Ο κύριο έλυσε τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά ο επόπτη για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον αναπληρωτή επόπτη προστασίας δεδομένων ε, που είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Η κυριαρχία των κρατών χωρών δεν είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να σεβαστούμε. Και δεύτερο, θα ήθελα κάποιες πληροφορίες για τη σχέση της ε, υπηρεσία, δηλαδή του επόπτη προστασίας δεδομένων με τις εθνικές αρχές. Για μένα δεν είναι σαφές οι χώρες μέλη πρέπει να είναι κυρίαρχες των πληροφοριών που διαθέτουν και εκείνες να αποφασίζουν σε ποιον θα στείλουν τις πληροφορίες και σε ποιον όχι. Και αν υπάρχει διαφορά μεταξύ μας δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Η Europol θα πρέπει να το σέβεται αυτό δεδομένου ότι είναι ο ενδιάμεσος ο κρίκος και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Πρέπει να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών ε, μελών, διαφορές μεταξύ των ε, συστημάτων που ισχύουν στι διάφορες χώρες και αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Βινιουρόφσκι για να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτές τις σημαντικές σε βάθο ερωτήσεις. Ξεκινήσουμε από την ε, γενική, το γενικό συμπέρασμα και αξιολόγηση ότι το νομικό σύστημα που θα πρέπει να διέπει την Europol σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και ισχυρό και αν υπάρξει ανάγκη να γίνουν επιπρόσθετες ε, εργασίες και διορθώσεις που θα είναι ενδεχομένω απαραίτητες σε κάποιο χρονικό σημείο. Όμως ήδη έχει συζητηθεί ο νέος κανονισμός για την προστασία δεδομένων στα ευρωπαϊκά όργανα. Όταν θα ξεκινήσουμε τις συζήτηση, λοιπόν, θα πρέπει αυτά, αυτά που θα αποφασιστούν να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς. Θα πρέπει να έχουμε ειδικέ λύσεις ε, για σώματα όπως η Europol. Λοιπόν, αποφάσισαν οι νομοθέτηση το σύστημα που ορίστηκε για την Europol πριν από τρία χρόνια είναι αρκετά ισχυρό και ίσως ακόμα και πιο κατάλληλο για τους ε, σκοπούς του, του οργανισμού. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σχέση με τις άλλες υπηρεσίε. Το ερώτημα του κύριου Βος, ναι, είναι ένα ισχυρό, ολοκληρωμένο σύστημα. Αν κάτι ένα πλαίσιο διορθώσεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα στην ε, διακριτική ευχαίρεια τη Europol. Οι πρακτικέ εργασίε είναι, είναι κομμάτι που πρέπει, με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η Europol, αλλά υπάρχει η ανάγκη να κοιτάξουμε τις νέες ε, λύσεις που προτείνουμε, ειδικά σε μια εποχή τόσο μεγάλων αλλαγών που έχουμε στα θέματα της ε, τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας. Η Europol ε, αλλάζει πολλά συστήματα πληροφορικής, όπως και άλλες υπηρεσίες αντίστοιχες. Άρα βοηθούμε να τους βοηθήσουμε να εφαρμόσουν αυτά τα συστήματα Υπάρχει και ένα άλλο θέμα με την ε, μεταφορά στις τρίτες χώρες. Είμαι βέβαιος ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες, οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Europol η ίδια ενδιαφέρεται πρωτίστως να λάβει τις πληροφορίες από τις τρίτες χώρες. Αυτό είναι κάτι για το οποίο είναι έτοιμη η Europol. είτε καλό είτε κακό, κάθε τέτοιου είδου συμφωνίε ε, συμπεριλαμβάνουν ε, αμοιβαιότητα. Μα δίνουν ε, τα δεδομένα, θα θέλουν να πάρουν και δεδομένα, να λάβουν δεδομένα. Ω βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε. Όπω είπα, είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε και την Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για να αξιολογήσει την κατάσταση. Ένα ερώτημα τέθηκε για την διαλειτουργικότητα αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του, αλλά συνδέεται ταυτόχρονα με τις καθημερινές εργασίες, ε, κυρίω της Γιώργου αλλά και Ιουλίζα. E Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στη διαβουλεύση την ε, διαλειτουργικότητα του Στρασβούργου την προηγούμενη εβδομάδα, στη συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου, όπου είχαμε συζητήσει με την Επιτροπή και με τους εκπροσώπους τη Ιουλίζα e και τους σκιώδεις συγητέ και τους συγητές του πακέτου διαλειτουργικότητας. Θυμάμαι, κάναμε λόγο για 6 και 7 βάσεις δεδομένων που, ε, στις οποίες υπάρχει διαλειτουργικότητα διαλειτουργικότητα. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό έδωξαν 40 βάσεις δεδομένων και πληροφορικά συστήματα που θα ε, λειτουργούν διαλειτουργικά στο ε, προσεχές μέλλον. Πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα γιατί αποφασίζουμε για τους πιο βασικούς κανόνες και αρχές για το προσεχές μέλλον. Ναι, εμπλεκόμαστε στη διαδικασία αυτή. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει προσκληθεί ε, στην ομάδα υψηλού πέδου για την διαλειτουργικότητα και συμμετείχαμε στις δραστηριότητες και σε ένα ε, σχέδιο που ε, προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Η συνεδρία στο Σασβούργο ήταν ε, λαμπρό παράδειγμα για την συνεργασία μας αυτή. Όσον αφορά τη χρήση των υποδομών της Europol από τα κράτη-μέλη, εμφανίστηκε και αυτό στις ερωτήσεις. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με, τις, ε, με τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Εποπτή Δεδομένων και των Εθνικών Αρχών Προστασία Δεδομένων. Και έχει σχέση και με την ε, συζήτηση για την διαλειτουργικότητα, γιατί η διαλειτουργικότητα δεν σημαίνει να περνάμε τα δεδομένα από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο επόμενο, αλλά είναι και το οργανωτικό κομμάτι της ε, διαδικασίας και η δυνατότητα του να, αποσπούμε, να μπορούμε να αποσπάσουμε και να εισάγουμε τα δεδομένα στα εθνικά συστήματα. Και φυσικά και σε εθνικό επίπεδο ε, τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να μοιραστούν όλα τα δεδομένα και αυτό με οδηγεί ε, στο θέμα της συνεργασίας με τους ε, αρχές, σε αρχές προστασίας δεδομένων. και ο Ευρωπαϊκό Επόπτη και τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται από τι εθνικέ του αρχές και προσπαθούμε να συζητήσουμε από κοινού όλα τα θέματα ε, που ε, είναι στο φάσμα των αρμοδιοτήτων μας και κυρίως αυτά που συνδέονται με την χρήση των υποδομών της Europol από τα κράτη-μέλη και ε, την μεταφορά των δεδομένων από, το εθνικ... από τις εθνικές αρχές στον Ευρωπαίο Επόπτη όσον αφορά την εφαρμογή στα κράτη-μέλη, το βασικό συντονιστικό σώμα είναι το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Προστασία των Δεδομένων, το οποίο αποτελείται από 28 εθνικές αρχές και από την Ευρωπαϊκό Προστασία των Δεδομένων και είναι το σώμα που έχει ευρύτερα καθήκοντα είναι υπεύθυνο για την εναρμόνιση ε, για το πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός στην πλησία δεδομένων στις, ε, στα κράτη-μέλη, αλλά και για το δεύτερο κομμάτι του πακέτου μεταρρύθμισης που έχει να κάνει με τις αρχές επιβολής ε, του νόμου. Όσον αφορά τη Frontex, ναι, Μα ρώτησαν αν είναι δυνατό να μεταφέρουμε ε, τα δεδομένα από την Europol στη Frontex και αντίστροφα και η Frontex ήδη έχει μεταφέρει τα δεδομένα στη Europol σε προσωπικά πακέτα δεδομένων. Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων από την Europol προς την Frontex που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για λειτουργικές ανάγκες δημιουργεί κάποια προβλήματα από νομικής πλευράς και θεωρήσαμε ότι δεν υπήρξε ε, επαρκής νομική βάση για να μπορέσει να γίνει αυτή η μεταφορά. Όταν λοιπόν ο Βος ρώτησε για, την, το κατά πόσο είναι πλήρως ολοκληρωμένο το σύστημα, είπα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σχετικό παράδειγμα. Έχουμε δύο υπηρεσίε που είναι πάρα πολύ καλέ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αλλά θα πρέπει να είναι βέβαιε ότι μπορούν να λειτουργήσουν ε, σύμφωνα με μια νομική βάση. Και αυτή τη στιγμή η μεταφορά των δεδομένων από τη Europol στη Frontex για λειτουργικού ε, σκοπού. Ε, για να γίνει αυτό μας λείπει η νομική βάση προτάθηκε λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βζιρόφσκι. Πριν περάσουμε στο επόμενο πάνελ, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια κι εγώ μετά από αυτά που είπε η κυρία Κινίτσι για την διαλειτουργικότητα και την προστασία δεδομένων, αλλά και όσον αφορά αυτό που ακούσαμε για την απουσία νομικής βάσης προκειμένου να υπάρξει μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στη Europol και την Frontex. Ε, λοιπόν, το πρόβλημα είναι μικρό σε σχέση με αυτό που θα σας πω τώρα. Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας συζητάμε για όργανα ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να πω ότι δεν μιλάμε μόνο για διαλειτουργική σχέση μόνο ανάμεσα στη Europol και τη Frontex για τα ΣΥΣ και τέτοια, αλλά και με την Interpol. Η Interpol απορρέει από τα Ηνωμένα Έθνη και είναι οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν οι περισσότερες χώρες του κόσμου. Πώς λοιπόν θα υπάρξει διαλειτουργικότητα των δικών μας μηχανισμών προστασίας δεδομένων με ένα τόσο ευρύ σώμα. Αυτό το δίνω ως τροφή για σκέψη. Γιατί υπάρχουν ήδη δύο νομοθετικές προτάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο κατάλληλος προπολογισμός και η κατάλληλη κατάρτιση για να μπορέσει να υπάρχει διαλειτουργικότητα ήδη σε κοινοτικό επίπεδο. Πώς θα τα καταφέρουμε όμως να έχουμε τέτοια διαλειτουργικότητα με την Ιντερπολ. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βιεβιρόφσκι για τα τόσο ενδιαφέροντα που μας είπατε και για ένα θέμα που μας απασχολεί τόσο πολύ αλλά και που προστατεύεται από ένα γερό σύστημα προστασίας που διαθέτει η Europol. Περνάμε τώρα στο επόμενο πάνελ εδώ θα ακούσουμε την Europol όσον αφορά τα οικονομικά εγκλήματα, ε, την νομοποίηση παράνομου χρήματος, για παράδειγμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Μάρτεν Ρέισενμπεκ, ο οποίος είναι εισαγγελέας, εθνικός εισαγγελέας, συντονιστής για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Είναι από τις κάτω χώρες. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Ντεμπόλε που είναι η εκτελεστική διευθύντρια της Europol. Και εκείνη θα παρέμβει. Και μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Πριν δώσω την προεδρία στο συνάδελφο Μπούχμαν, επιτρέψτε μου να πω ότι η νομοποίηση παράνομου χρήματος, η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος είναι πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία συνδέονται και επηρεάζουν και άλλους τομείς του εγκλήματος. Το κοινό έγκλημα, είτε πρόκειται για ναρκωτικά, είτε πρόκειται για ε, σωματεμπορία, λαθρεμπόριο κλπ. Υπενθυμίζω ότι ο τέος διευθυντής της Europol πολλές φορές μας είχε πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για την ε, Κοινή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Εξού και με ιδιαίτερη χαρά, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρουσιάζω τον κύριο Μάρτεν Ρέισενμπεκ, ο οποίο, όπω είπαμε, είναι εθνικό αγγελέα συντονιστή για την καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία από τι κάτω χώρε και θα μα παρουσιάσει το πρόγραμμα τη δικιά του χώρα, τη Ολλανδία δηλαδή, όπου συνεργάζονται η αστυνομία, οι εισαγγελεί και οι τέσσερι μεγαλύτερε τράπεζε τη χώρα προκειμένου να εξετάζουν οικονομικά στοιχεία και δεδομένα και να αποφεύγονται τρομοκρατικές ενέργειες. Στη συνέχεια θα ακούσουμε, είναι εδώ, η κυρία Ντεμπόλε που είναι εκτελεστική διευθύντρια. Και σταματάω εδώ. Σοπαίνω. Γιατί νομίζω ότι θα προεδρεύσει καλύτερο ο συνάδελφος Μπούχμαν. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, Ριζεμπέκ, ο λόγος σε uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην πρόληψη τρομοκρατίας και έρευνα για την τρομοκρατία είναι κρίσιμη σημασία ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και πώς χρηματοδοτείται η τρομοκρατία. Στην Ολλανδία ο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα συνεργάζονται. Ερευνούν κατά πόσο η συνεργασία του μπορεί να συμβάλλει σε μια προσέγγιση σωστή. Και μεγάλη τιμή για μένα να μοιραστώ μαζί σα τι γενικέ γραμμέ και τα αποτελέσματα τη Ολλανδική προσέγγιση και τη ομάδα κρούση για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Είναι συνεργασία ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Οι τέσσερι μεγάλε εθνικέ τράπεζε και μια ασφαλιστική εταιρεία, η FIU, η Εθνική Αστυνομία, ε, οι, υπηρεσίες εφορίας και οι υπηρεσίες ένωσαν τις δυνάμεις για πρόληψη και έρευνα της χρηματοδοτήσεως των τρομοκρατών. Στις έρευνές μας επιθυμούμε διακαώς να διαρευνήσουμε τις τάσεις που υπάρχουν, όπως νέες μέθοδοι πληρωμής. Σε κάθε έρευνα που κάνουμε, είτε έρευνα κατοικίας ή ηλεκτρονικών συσκευών, ψάχνουμε για στοιχεία στοιχεία που θα μας δείξουν καινοτόμου τρόπους χρηματοδοτήσεως των τρομοκρατών. Προς έκπληξη μας δεν βρίσκουμε πολλά τέτοια νέα φαινόμενα. Και δεν λέω ότι δεν χρησιμοποιούνται νέε μέθοδοι πληρωμών σε μεγάλη κλίμακα, αλλά παρά τις προσπάθειές μας δεν έχουμε εντοπίσει την υποδομή αυτή μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η τρομοκρατία. Προφανώς θα εστιαστούμε πάνω σε νέε μεθόδου πληρωμή, να παρακολουθούμε αν είναι ευάλωτε και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση τρομοκρατία. Εν το μεταξύ όμω, βλέπουμε πολλέ παραδοσιακέ τακτικέ χρηματοδοτήσεω. Μικροχρηματοδότηση, Φερρυπίν, μέσω του συνηθισμένου τραπεζικού συστήματο, χρήση εμβασμάτων συνδυαζόμενη με διμεσάζοντε για να κρύβονται οι προορισμοί οι τρομοκρατικοί και άλλου είδου ε, και που δεν έχουν τη σωστή άδεια. Είναι πολύ δύσκολο για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να εντοπίσουν τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών μέσω ε, της συνηθισμένου ελέγχου των πελατών και διακίνησης χρημάτων. Και αυτό για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν πολλοί αποτελεσματικοί τρόποι χρηματοδότησης τρομοκρατών που έχουν αναπτυχθεί και τυπολογίες. Και δεν πρέπει να στεζόμεθα μόνο στην προέλευση των χρημάτων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατία, που μπορεί να είναι νόμιμη πηγή, αλλά πρέπει να βλέπουμε και ποιο είναι ο προορισμό. Όσο απομακρύνεσαι από τον τελικό προορισμό των τρομοκρατών, τόσο πιο δύσκολο είναι να κατανοήσει τι ψάχνει να βρει. Κυρίω όσον αφορά σχετικά μικρά ποσά, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Εν τω μεταξύ, τα διεθνή πρότυπα και εθνικέ νομοθεσίε απαιτούν από τα χρηματοσυντικά μα ιδρύματα να εντοπίσουν αυτέ τι συναλλαγέ και του τρομοκράτες που εμπλέκονται στι συναλλαγές αυτέ. Λαμβάνουμε κάσες ε, εκθέσεις περί υπόπτων συναλλαγών υψηλού που έχουν εντοπιστεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Το SDR ε, ήταν πολύ σημαντικό για τις έρευνές μας. Πολλές από τις έρευνές μας ξεκίνησαν βάσει τέτοιων STRs. Και έτσι η παρακολούθηση συναλλαγών των κανονικών πελατών από τον χρηματοδοτικό τομέα δίνει στις δυνάμεις επιβολής του νόμου καλές πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεχώς προσπαθούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών που καταναλώνουν για τον εντοπισμό της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν σημαντικές πληροφορίες στη διάθεσή τους. Προσωπικά στοιχεία και σχετικά ε, στοιχεία επαφών ε, με ανθρώπους που θεωρούνται ότι είναι τρομοκράτες. Όπως ήδη ανέφερα, τα χρηματοστικά ιδρύματα υπέχουν νομική υποχρέωση να εντοπίσουν αυτούς τους ανθρώπους εντός του πελατολογίου τους και να αναφέρουν και να καταγγέλουν ασυνήθιστες συναλλαγές στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται τρομοκράτες οι υπηρεσίε ιδιοκτικέ και οι δυνάμει επιβολή του νόμου έχουν την άποψη ότι κατεπηγόντω απαιτείται τα χρηματοδοτικά ιδρύματα πραγματικά να προβαίνουν σε αυτού του ελέγχου και τι καταγγελίε. Αν θέλουμε όμω να βρουν τι πληροφορίε, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τι ευκαιρίε που έχουμε στα νομικά μα πλαίσια ε, να του δώσουμε τι πληροφορίε που απαιτούνται. Και αυτό ξεκινήσαμε σε ένα πιλωτικό μα ε, πρόγραμμα η ομάδα κρούση για την καταπέσταση τρομοκρατίας είναι οργανωμένη μέσα στο ε, στο κέντρο που εσχαρείται με τα δημοσιονομικά. Συνεργάζεται, είναι συνεργασία αρχών που έχουν υποπτικό έλεγχο, διοκτικές αρχές και ερευνητικά καθήκοντα. Ιδρύθηκε το 1997 για να ενισχύσουμε την ακαιρεότητα του χρηματοστοτικού τομέα. Κινούμενοι εντός του νόμου, χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πληροφορίες και τη σχετική νομοθεσία και συντονιζόμενη με τις διοκτικές υπηρεσίες, η αστυνομία μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες πολύ σημαντικές με τους ιδιωτικούς εταίρους αυτής, περί τρομοκρατών και περί εκείνων που τους διευκολύνουν και που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Αυτές οι πληροφορίες ερευνώνται περαιτέρω από τους ιδιωτικούς μας εταίρους και ασυνήθιστες συναλλαγές καταγγέλλονται και επιστρέφονται στις αρμόδιες αρχές. Το FIU αναλύει τις ασυνήθιστες συναλλαγές και παρέχει στις νομικές υπηρεσίες σχετικές εκθέσεις περιπόπτων συναλλαγών προς έρευνα και προς εξυχνίαση. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες περί ασυνηθίστων συναλλαγών που έχουν εντοπίσει με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ε, το οποίο ε, εξετάζει ε, την όλη συναλλαγή του ομολόγου. Τι ο τρόπος τα χρηματοστικά ιδρύματα είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν ενδεχόμενα δίκτυα τρομοκρατών και να εντοπίσουν και να αναφέρουν ενδεχόμενες άλλες ασυνήθιστες συναλλαγές οι οποίες εμπλέκονται και να καταγγέλουν αυτές στις αρμόδιες αρχές. Τι ούτω τρόπος, σε κάποιες περιστάσεις, διμερείς πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ ιδιωτικών εταίρων είναι κάτι εφικτό εντός της Task Force. Όμως, πολυμερής ανταλλαγή πληροφοριών θα ήταν πολύ αποτελεσματικότερη εν αυτή περίπτωση και ότι το νομικό μας πλαίσιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο είναι κάτι που θεωρείται ως εμπόδιο. Στην Task Force, λοιπόν, οι αναλυτές των ιδιωτικών μας εταίρων εργάζονται στο ίδιο γραφείο όπως και οι αναλυτές των αστυνομικών αρχών και το FIU για να μειώσουμε τον αντίκτυπο τη ιδιωτικότητα των στοιχείων και τη σύμπραξη αυτή, η Task Force είναι ένα κλειστό κουτί, όπω αποκαλείται. Οι πληροφορίε που ανταλλάσσονται μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών δεν μπορεί να φύγει από την ομάδα κρούση, από την Task Force. Δεν επιτρέπεται ο αναλυτής του ιδιωτικού τομέα να σώσει τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων της εταιρεία για την οποία εργάζεται ή να μοιραστεί τις πληροφορίες αυτές με έναν συνάδελφο ο οποίος δεν εργάζεται εντός της Task Force. Μόνο οι συνήθιστες συναλλαγές οι οποίες έχουν αναφερθεί στο FIU γίνονται ορατές στο υπόλοιπο τμήμα συμμόρφωσης εταιρείας. Και αυτές είναι συναλλαγές που θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί και να καταγγελθεί ούτως ή άλλως. Χρειάζεται μεγάλο θάρρος και από το δημόσιο και τον ιδιωτικό εταίρο να συνεργαστούν τούτο τρόπος. Αν μοιράζεται κανείς πληροφορίες με άλλους, είτε στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ο κίνδυνος αποκάλυψης των πληροφοριών αυτών αυξάνεται. Όμως το επίπεδο εμπιστοσύνης σε αυτή την task force είναι ύψιστο και δεν έχει παραβιαστεί που δεν είναι. Τα προσωρινά αποτελέσματα του πιλωτικού προγράμματος καταδεικνύουν ότι αυτή η σύμπραξη ε, απέδειξε ότι δίνει ποιότητα, ποσότητα ε, και έδωσε σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την καταγγελία υπόπτων συναλλαγών. Το πρώτο έτος οι αστυνομικοί μοιράστηκαν 15 υποθέσεις με τους ιδιωτικούς εταίρους και αυτό οδήγησε στην εξυχνίαση και καταγγελία πάνω από 300, ε, συναλλαγών. 64% από αυτές τις συναλλαγές ε, δηλώθηκαν ύποπτες από το FIU και διαβιβάστηκαν στις αστυνομικέ δυνάμεις. Κατά μέσο όρο περίπου 10% όλων των ασυνηθίστων συναλλαγών δηλώνονται ύποπτες στην Ολλανδία. Λόγω του υψηλού, υψηλής προτεραιότητας των υποθέσεων που χειρίζεται το Task Force, τα SDR που απορρέουν από εκεί χρησιμοποιούνται άμεσα σχεδόν από τις αστυνομικέ υπηρεσίες. Πέραν αυτού, οι εταίροι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μοιράζονται βέλτιστε πρακτικέ και μεθόδου ε, εντό τη Task Force για την έρευνα για την καταπληκτική τη τρομοκρατία. Τέτοια αποτελεσματική. Είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τυπολογίε που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτε και γι' αυτό απαιτείται επιγόντω ανταλλαγή πληροφοριών με τον τρόπο που δοκιμάζουμε. Ψάχνουμε να βρούμε νέου καινοτόμου τρόπου για να εντοπίζουμε την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση τρομοκρατών εγκαίρω μέσω μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Είμαι υπερήφανο, διότι οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί εταίροι συνεργάζονται επικοδομητικότατα. Παραδεχόμενοι το καθήκον και τι ευθύνε του καθενό, έχουμε κοινού στόχου. Η του χρηματοδοτικού ε, τομέα και έρευνα και η εξυχνίαση τρομοκρατία και χρηματοδότηση τρομοκρατία είναι οι στόχοι μα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και με τα χαρά να απαντήσω ερωτήσει σα. Σας ευχαριστώ κύριε Ιζεμπέκ για την ε, παρουσίασή σας. Θα προσκαλέσω την κυρία Ντεμπόλ να πάρει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Ντίας μερα, κύριε Μπούχμαν, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα που είναι η εγκληματικότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πολλές ε, ανακτήσεις επιτεύχθηκαν ε, το 2018. Ήταν μία από τις κύριες προτεραιότητές μας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ήταν μία από τις προτεραιότητες της Europol. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε τους εγκληματίες συστηματικά. Πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εγκληματικές ε, χρηματοπιστωτικές ροές. Σήμερα θα σας εξηγήσω ποιος είναι ο ρόλος της Europol στην καταπολέμηση του χρηματοπιστωτικού εγκλήματος και θα σας ε, πω και ποιο είναι το μέλλον. Προηγουμένως όμως θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις τάσεις και τις εξελίξεις που βλέπουμε στο θέμα της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Ποιες είναι οι τάσεις. Το έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι σε μερικές περιοχές τα κέρδη από το λαθρεμπόριο συνθετικών ναρκωτικών είναι πάνω από 20 δισεκατομμύρια ετησίως. Η νομοποίηση λοιπόν παράνομου χρήματο είναι μια πολύ μεγάλη ανησυχία για μα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει τα κέρδη αυτά οι εγκληματίε να τα νομιμοποιούν με κάποιο τρόπο. Και ακριβώ αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Η νομοποίηση λοιπόν του εγκληματικού αυτού χρήματο ε, αποτελεί και αντικείμενο πολλών συγκεκριμένων δράσεων. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένε ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα σωρό εγκληματικέ δραστηριότητες ακριβώς για την νομοποίηση του παράνομου χρήματος. Και μερικές φορέ υπάρχουν και συνδέσεις με τρομοκρατικέ ομάδες. Αυτές οι ομάδες είναι ιδιαίτερα καλά και είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα με πολύ περίπλοκε υποθέσει βασίζονται στη χρήση του ρευστού, στην ε, κατάχρηση εταιρικών δομών και στην εκμετάλλευση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των επενδυτικών αγορών. Για παράδειγμα, είχαμε την Κοντίνη Σανταλουτσία, την πρόσφατη δηλαδή δράση μας, η οποία οδήγησε στην Ιταλική Καμόρα τελικά η ομάδα κατάφερε να νομιμοποιήσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ την εβδομάδα πάνω από 250 εκατομμύρια τελικά νομοποιήθηκαν μέσω ενός περίπλοκου συστήματος χρησιμοποιώντας couriers ρευστού με ε, καταχρήσεις και χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι εγκληματίες βασίζονταν σε παραδοσιακές μεθόδους νομοποίησης παράνομου χρήματο. Όμως υπάρχουν και αναδύονται και νέες μέθοδοι. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη δράση μας Dryer, εκεί διαπιστώσαμε ότι παρεμβαίνει και το, παρεμβαίνουν και τα κρυπτονομίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται από εγκληματικές ομάδες που παράγουν συνθετικά ναρκωτικά και τα κυκλοφορούν. Η νομοποίηση παράνομου χρήματο μέσω κρυπτονομισμάτων είναι κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο. Υπάρχουν νέε μέθοδοι πληρωμή που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα όπω οι παραδοσιακέ και έτσι επιτρέπουν να γίνονται εύκολα διασυνοριακά συναλλαγέ που δεν εντοπίζονται από τα συστήματα ελέγχου και αναφοράς που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι υπάρχουν νέες ευκαιρίες για την νομοποίηση παράνομου χρήματος, κάτι το οποίο αποκτά όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα μεταξύ των εγκληματιών. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε νέες μεθόδους, σε νέους μηχανισμούς για να μπορούμε να εντοπίζουμε αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Τι κάνει η Europol τώρα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Έχουμε ένα τμήμα πληροφοριών, για αυτό ακριβώς ε, το θέμα, για την καταπολέμηση λοιπόν του, κλιματικού, του οικονομικού εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχειρησιακά πρώτα απ' όλα. Το τμήμα μας στηρίζει τις έρευνες και την ανάκτηση κεφαλαίων στις διάφορες χώρες μέλη. Επίσης, προσφέρουμε και πληροφορίες για να στηρίξουμε έρευνες που γίνονται σε άλλες περιπτώσεις εγκλημάτων, λαθρεμπόρων ναρκωτικών, απάτες, τρομοκρατία κτλ είναι κεντρικό στοιχείο η καταπολέμηση του, του οικονομικού εγκλήματος στη Europol. Ελέγχουμε λοιπόν μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε, ύποπτες συναλλαγές ας πούμε από διάφορα FIUs ή από κατασχέσεις ρευστού στα τελωνία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια πλήρη εικόνα ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνδέσεις ανάμεσα στις διάφορες μορφές ε, οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτή η στήριξη ε, είναι κάτι που προσφέρουν και οι χώρες και ζητούν μάλλον οι χώρες όλο και περισσότερο. Το 2017 η ανταλλαγή πληροφοριών για ανάκτηση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 81% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο αριθμός των οικονομικών ε, ερευνών που στηρίξαμε αυξήθηκε κατά 110% και η Europol σήμερα στηρίζει 221 περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητες, 13 δράσεις επίσης στηρίχθηκαν το πρώτο εξάμεινο του 2018 από μας σε σχέση με 8 το αντίστοιχο διάστημα του 2017. 257 συλλήψεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που είναι αντίστοιχο 37 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, εμείς φιλοξενήσαμε και το κεντρικό σύστημα υπολογιστών των FIU για ανάπτυξη παρετέρω δραστηριοτήτων όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε στρατηγικό επίπεδο. Η Europol έχει δεσμευτεί να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των ε, πλευρών που φροντίζουν για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Στηρίζουμε λοιπόν ε, διάφορα επαγγελματικά δίκτυα όπως είναι το Recolt, την πλατφόρμα ή την τριμερή ομάδα εργασίας για τα ψηφιακά νομίσματα. Έτσι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης των οικονομικών εγκλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ποιο είναι το μέλλον ε, των ε, οικονομικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες, η πραγματογνωμοσύνη που διαθέτει η Europol είναι ε, κεντρικό στοιχείο όσον αφορά την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Έτσι μπορούμε να προβούμε σε συστάσει για το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Έγινε μια έρευνα από την Europol που έδειξε ότι μόνο 1% των ε, εγκληματικών ε, διαδικασιών ε, που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγουν σε κατάσχεση. Και σε 10 χρόνια μόνο 10% των ύποπτων συναλλαγών και με τον ιδιωτικό τομέα τελικά κατέληξαν σε διερεύνηση. Υπάρχουν κάποιες ακαμψίες όσον αφορά τις υποδομές και αυτό ευθύνεται για τα κακά αποτελέσματα που έχουμε. Πάντως η ομάδα πληροφοριών για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος έχει, παίρνει κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο αναφορές για ύποπτες συναλλαγές. Και οι αναφορές αυτές ως ε, επιτοπλίστων δεν συνοδεύονται από πληροφορίες και τελικά χάνονται μέσα στον όγκο των ε, πληροφοριών. Έπειτα, εμποδίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών μερικές φορές. Δεν υπάρχει δηλαδή συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων οικονομικών πληροφοριών ή και για την ανταλλαγή με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα FIUs μπορεί να βοηθήσει να ενισχύσουμε στις έρευνές τους τις αρχές που ερευνούν οικονομικά εγκλήματα. Πρέπει δηλαδή αυτούς τους περιορισμούς να τους ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, γιατί οι οικονομικές πληροφορίες αποτελούν ο ακρογωνίο λίθο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να βρούμε το οικονομικό έγκλημα και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να καταργηθούν τα εμπόδια και να υιοθετήσουμε μια πιο σωστή προσέγγιση. Στην Europol διαθέτουμε τη γνώση και βοηθούμε και τις εθνικές αρχές. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή της γνώσης μπορεί να βοηθήσει και τις εθνικές αρχές να εντοπίσουν καλύτερα τις ύποπτες συναλλαγές. Με αυτό ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2017 με ένα πιλωτικό πρόγραμμα όσον αφορά την εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα, όπου διεθνείς τράπεζες και διάφορες εθνικές αρχές συμμετέχουν. Τέλος, θα έλεγα ότι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος πρέπει να διευκολύνουμε τις έρευνες και την ε, ανάκτηση κεφαλαίου μέσω ερευνών και να ενισχύσουμε τη νομική, τη νομική υποδομή που διαθέτουμε και τους μηχανισμούς, όπως επίσης να υπάρξει και περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ εταίρων. Γι' αυτό και είναι φρόσδεξη η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα οδηγία όσον αφορά τη χρήση των οικονομικών πληροφοριών και κυρίως μας αρέσει η πρόταση που λέει ότι η Europol θα έχει έμεσα πρόσβαση σε μητρό τραπεζικών λογαριασμών και ότι θα μπορεί να ζητάει πληροφορίες από την ε, Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών. Το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή τέτοια ομάδα οικονομικών πληροφοριών που να συντονίζει το έργο των εθνικών FIUs. Το βασικό στοιχείο θα ήταν πρόσβαση σε όλες τις διασυνοριακές συναλλαγές αλλά και στις κατασχέσεις ρευστού οι δηλώσεις ρευστού που είναι στη διάθεση των τελωνιακών αρχών. Έτσι η Europol θα μπορούσε να στηρίξει καλύτερα τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ντεμπόλ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με το διάλογο και ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος Γκρέχ από τη Μάλτα. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ αγαπητοί ε, συνάδελφοι, καθώς ε, εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη τόσο ραγδαία, θα πρέπει να καταβάλουμε τις καλύτερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε ε, το οργανωμένο έγκλημα και το κυβερνό έγκλημα που μπορεί να επηρεάσει τις ζωές των πολιτών, τις οικονομίες μας και τις υποδομές. του κυβερνό έγκλημα έχει μεγαλύτερη διάχυση καθώς η χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι το internet banking και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξαπλωθεί επιπλέον. Είναι προφανές ότι ο ρυθμός ε, ε, της εξέλιξης ε, της τεχνολογίας είναι πολύ πιο γρήγορος από την αλλαγή στην νομοθεσία. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πολίτες δεν είναι καλυμμένοι από την απαραίτητη και κατάλληλη νομοθεσία. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε λοιπόν περαιτέρω τους πολίτες μας, τους κινδύνους που καιροφυλακτούν. Επίσης έχουμε απειλές τρομοκρατίας και αστάθειας στις γειτονικέ χώρες όπως είναι η Λιβύη ε, και η Συρία. Αυτή η αστάθεια στη γειτονιά της Ευρώπης πυροδοτεί ε, εγκληματικές δραστηριότητες όπως είναι η εμπορία ανθρώπων, ε, η οποία συνδέεται και με την παράνομη μετανάστευση. Ε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ε, ε, εκατομμύρια, ε, ευρώ τα οποία εισραίουν παράνομα στο οικονομικό μας σύστημα. Εν ώψη λοιπόν αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο η Europol να κτίσει τις ικανότητες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές ε, τις ε, προκλήσεις και στις ε, χώρες μας αλλά και στις γειτονικέ χώρες. Θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου ε, για το πολιτές πρόγραμμα της Europol 2009-2021 και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταστήσουμε, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στις χώρες μας. Εύχομαι να συνεχίσει τις επιτυχίες της η Europol και να μπορέσει να λύσει ε, τα αποτελέσματα από το παρελθόν για να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει τα μαθήματα από το παρελθόν. Επίσης ε, ε, ελπίζω να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι αυτή η ομάδα για να μπορέσει η Ένωση μας να έχει την ασφαλή και την ευημέρεια που της αρμόζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Κιδιός από την Κύπρο. Γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την λεπτομερή ενημέρωση. Κυρία Ντεπόλ, ε, έχετε ήδη απαντήσει πολλά από τα ερωτήματα τα οποία ε, έτσι σχεδιάζαμε να υποβάλουμε. Ωστόσο, ε, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση την οποία κάνατε για την αυξανόμενη χρήση των κρυπτονομισμάτων. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν, ε, εάν είναι η Europol και οι εθνικές αρχές σε θέση να εντοπίζουν αποτελεσματικά την προέλευση των παράνομων πράξεων που τελούνται σε κρυπτονομισμά και πώς μπορεί να εμπλακεί πιο ενεργά ο ιδιωτικός ε, τομέας σε αυτές τις ε, έρευνες οι οποίες ενδεχομένως να γίνονται. Όσον αφορά το ζήτημα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ε, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν διευκολύνει η Europol την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών και αν έχετε κάποια στατιστικά, αν υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στον τομέα της παράνομης διακίνησης, της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι η κυρία Γκόμες από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Συμμετείχα στο σχεδιασμό του τέταρτου και της τέταρτης και πέμπτης ε, ε ομάδας για την οδηγία για την καταπολέμηση της ομοιπήμησης των εσόδων. Ε, με ικανοποίησαν αυτά που έξω από τους ομιλητές και ειδικά τις πληροφορίες που είχαμε από το Αθηνικά Κοινοβούλιο ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει προτείνει στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το πέμπτο, την πέμπτη πολιτική οδηγία για την καταπολέμηση του ξέπλυμα του χρήματος, να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό FIU για να διασφαλίσουμε ότι θα μοιραζόμαστε τις πληροφορίες όχι μόνο σε επίπεδο FIU και να μην εμποδίζουμε τις ε, εταιρικές σχέσεις οι οποίες Υπάρχουν. Αυτό όμως το αρνήθηκαν τα κράτη-μέλη από το Συμβούλιο. Είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζετε. Θα πρέπει να, γνω... να ρωτήσετε τις κυβερνήσει γιατί το αρνήθηκαν. Προφανώ δεν ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση του ξεπλήματο του χρήματο. Και έχοντα εργαστεί εντατικά σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι κάποιες κυβερνήσει διευκολύνουν την νομιμοποίηση παράνομων, παράνομου χρήματος. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ότι αυτοί που διαβουλεύονται δεν είναι άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση του εγκλήματο, αλλά είναι άτομα του Υπουργείου Οικονομικών που θέλουν να διευκολύνουν την ομοποίηση παράνομων εσόδων. και αδιαφορούν για την καταπολέμηση του εγκλήματος επίσης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε ένα πρόσφατο σημείο της σχετικής οδηγίας για την καταπολέμηση των παράνομων εσόδων ε, που πέρασε στο Κοινοβούλιο μετά τέτοια διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο κτλ. και αφορά το ποινικό δικαίο, προτείνει το Κοινοβούλιο ότι θα υπάρξουν δυσμενείς εξελίξεις για αυτούς που μπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες γιατί θα είναι άτομα από τον πολιτικό χώρο που θα εκτεθούν. Εσείς, εγώ, άτομα στις κυβερνήσεις που διευκολύνουν τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτό, λοιπόν, απορρίφθηκε από κάποιες κυβερνήσεις και μπορώ να σας πω ποιες είναι αυτές που το αποφεύγουν, το εμποδίζουν. Είναι κάτι που με εξοργίζει η Επιτροπή. Άλλο παράδειγμα. Εδώ και ένα χρόνο έχει προτείνει να εξαλείψει τα παρθυράκια στο σύστημα VIT που δίνει δυνατότητα στο οργανωμένο έγκλημα και τις τρομοκρατικές ε, οργανώσεις όπως είναι η Αλκέιντα να εκθέσει ε, το σύστημα VAT μέσω μιας απάτης καρουζέλ. Τίποτα δεν έγινε τελικά. Η Επιτροπή υπολογίζει ότι αυτό αντιστοιχεί σε 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μπορείτε να το αναλύσετε 50 δισεκατομμύρια. Είναι το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Άρα οι κυβερνήσει μας θέλουν πραγματικά να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα του χρήματο και θα ολοκληρώσω. Με μία ερώτηση μπορούσα να συνεχίσω, αλλά θα ολοκληρώσω και θα ρωτήσω. Γίνανε πολλέ αναφορέ στο κρυπτονόμισμα. για ανώνυμους για την ε, κατάργηση των ανώνυμων μετόχων και ότι θα πρέπει οι εταιρείε ουσιαστικά να ε, κατονομάσουν τους δικαιούχους και όχι μόνο αυτού που είναι εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτού που δραστηριοποιούνται και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέλουν οι κυβερνήσει μα ήταν πολύ εύκολο να γίνει, αλλά δεν το θέλουν. Άρα το ερώτημά μου αφορά έναν άλλον τομέα που είναι πολύ δύσκολο να ρυθμιστεί και βλέπουμε ότι ήδη κάποια κράτη-μέλη ε, είναι κόμβοι για κρυπτονομίσματα και για την τεχνολογία blockchain και η ερώτησή μου σε εσά είναι ότι κάποιοι προτείνουν οι τεχνολογίες blockchain είναι πολύ σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι αυτό αποτελεί προπαγάνδα για να επιτραπεί η ανάπτυξη του κρυπτονομίσματος. Όπως ήδη τονίζετε, τονιστεί, υπάρχουν νέα εργαλεία τα οποία τα, ε, προσπαθούν να τα εξελίξουν ε, οι, τρομοκρατα... οι, τρομο... οι εγκληματικές οργανώσεις. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος ε, στον αντιπρόσωπο από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματο, δηλαδή η νομοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που αφορά δημόσιου λειτουργού και δημόσιου υπαλλήλου με την ευρία έννοια, απασχολεί τις αρχές όλων των κρατών μελών, αφού προστατεύει τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, υφυπουργοί κλπ. απέκτησαν χρήματα με παράνομες πράξεις που έγιναν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επευκαιρία ή και με αφορμή αυτά. Τα εγκλήματα αυτά συνήθως είναι η παράβαση καθήκοντος, η απιστία περί την υπηρεσία και η δωροδοκία ή δωροληψία του δημοσίου προσώπου, κλπ. Ε, με βάση το Σύνταγμα της Ελλάδας και το, δικαιοπολιτικό, το Σύνταγμα της Ελλάδας και το δικαιοπολιτικό της σύστημα, οι πράξεις των προσώπων αυτών υπάγονται σε βραχυχρόνιες προθεσμίες παραγραφής, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα αυτά, αν και προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες, να μην τιμωρούνται λόγω παραγραφής των εγκλημάτων αυτών, σε αρκετές περιπτώσεις. Ήδη, οι περιπτώσεις αυτές καταχρηστικής και παράνομης άσκησης των αρμοδιοτήτων δημοσίων λειτουργών του παρελθόντος εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα θέματα η Ελλάδα τα αντιμετωπίζει γενικά με τις δικές της δυνάμεις. Υπάρχει ουσιαστική συνεργασία του Γεροπόλ και των κρατών μελών και σε ποιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού του είδους διαφοράς. Ευχαριστώ. Thank σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι από την Εστονία. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομα. Είναι ο κύριος Εκ. Äh, äh, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά που λέγαμε τη συζήτηση και κυρίως αυτά που είπε ο Ολλανδός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της Europol, εγώ ενδιαφέρομαι για ένα άλλο θέμα, για το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και θεσμών που εργάζονται στον τομέα του ξεπλήματος ε, χρήματος. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη δική τους εμπειρία, έχουν τις δικές τους διαδικασίες και είναι, αρκετά, είναι κλειστά κυκλώματα το ΣΥΠΗΝ αυτές οι διαδικασίες. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε περιπτώσεις σαφώς ποινικών ε, δραστηριοτήτων. Σε άλλες περιπτώσεις οι πληροφορίες και τα δεδομένα ε, παρακρατούνται απομονωμένα. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση στην οποία οι ποινικέ δραστηριότητε δεν εντοπίζονται σαν αποτέλεσμα αυτό. Με ενδιαφέρει το πείραμα το Ολλανδικό και η εμπειρία η Ολλανδική. Ποια είναι η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος, ε, αντιμετώπιση του, του θέματος του ξεπλήματος χρήματος και των Ολλανδικών αρχών. Ε, μια ερώτηση προς τη Europol. Ποια είναι η άποψη της Europol. Αξίζει να αυξηθεί η ανταλλαγή στοιχείων. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σε περιπτώσεις ύποπτων ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Επομένω, εκπρόσωπο από το Ευρωκοινοβούλιο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλω να συγχαρώ την κυρία Μπόλε για την παρουσίαση της, πολύ ενδιαφέρουσε τι παρουσιάσεις και αξίζει πάντα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονε. Καταλαβαίνω και ολλανδικά και αυτό το κάνει όλα πιο απλά, δεν χρειάζεται δηλαδή μετάφραση. Όσον αφορά πρώτα απ' όλα τη συνεργασία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Όταν υπάρχει επιτυχία είναι ακριβώς επειδή υπάρχει καλή συνεργασία. Ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Αυτή η συνεργασία είναι κλειδί, η βάση της επιτυχίας. Από εκεί και πέρα βέβαια αποδεικνύεται δύσκολο πολλές φορές γιατί εσείς πρέπει να δουλέψετε με τα μέσα που διαθέτετε. Έχετε νομικές δυνατότητες, αλλά έχετε και νομικούς περιορισμούς. Υπάρχει θέμα κυριαρχίας, υπάρχει θέμα εντολής που πρέπει να σέβεστε. Και πρέπει βέβαια να συλλάβετε όσο γίνεται περισσότερους εγκληματίες και να καταλήξουν στη φυλακή. Καταλαβαίνω λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το έργο σας. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως επίσης είναι κατά πόσο ε, αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συμβαίνει και στο λεγόμενο σκοτεινό δίκτυο, dark web. Κατά πόσο δηλαδή εσείς καταλαβαίνετε τι γίνεται με τα κρυπτονομίσματα, πώς κυκλοφορούν, πόσο. Και τέλος την κυρία Ντεμπόλε θέλει να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε σε ένα εκατομμύριο αναφορές από τα FIUs. Ίσως να μην σας άκουσα καλά, αλλά επρόκειτο για κανονικές συναλλαγές ή για ύποπτες συναλλαγές. Σε εθνικό επίπεδο τα FIUs δουλεύουν βάσει δικτών, έτσι δεν είναι. Και έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια διεθνής έρευνα. Αλλά πρόκειται για κανονικές συναλλαγές ή όχι. Οι υποθέτω ύποπτες. Είπατε ότι είναι πολύ δύσκολο σε επίπεδο Europol να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών επαρκής. Υπάρχουν κάποιοι που ζητούν ένα ευρωπαϊκό FIU, είπατε επίσης. Δεν ξέρω αν αυτό το θέλω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα της Europol όπου να συμμετέχουν οι εθνικές αρχές, τα εθνικά FIUs και να μπορούν υπό την αιγίδα της Europol να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες τους. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα τέτοιο μηχανισμός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Επόμενος από το Ευρωκοινοβούλιο, η κυρία Τσίνετζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους φιλοξενούμενους μας για τις παρουσιάσεις τους. Ήταν πλήρεις, επίκαιρες και πραγματικά συμφωνούσα με αυτά που παρουσίασαν. Ήδη δόθηκαν απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να θέσω και έγιναν και πολλέ άλλε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τους προλαλήσαντε συναδέλφου. Πιστεύω και λόγω τη επαγγελματική μου, του επαγγελματικού παρελθόντος, ε, εγώ προέρχομαι από την Ιταλία. Εκεί η συνεργασία απεκαλύφθη βασικό όπλο στην ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπατε, αυτό που είπε η κυρία Ντεμπόλ, αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησε είπε ότι πρέπει να πλήξουμε την εγκληματικότητα εκεί που κάνει το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή στα χρηματοστατικά τους ε, και τα οικονομικά τους συμφέροντα. Διότι αυτή είναι και η ιστορία της χώρας μου. Εξετίμησα πάρα πολύ αυτό που παρουσίασε ο κ. Σεμπέργκ, Ζητώ συγγνώμη για, την, για το όνομά σας όπως το προφέρω, διότι ανταποκρίνεται σε αυτό στην εμπειρία της Ιταλίας και δείχνει πως αυτή η συνεργασία πραγματικά είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για να αντιταχθούμε στα εγκλήματα τα οικονομικά. Τα οικονομικά εγκλήματα διαδίδονται όλο και περισσότερο και συναρτήσει της χρήσεως ε, των πληροφορικών μέσων από πλευράς των εγκληματιών. Μπορούν να μεταφέρουν εύκολα χρήμα μέσω της χρήσεως κρυπτονομισμάτων κλπ. μέσω μιας σειράς μηχανισμών και πάνω σε αυτό διερωτώ αυτή είναι η ερώτησή μου που θέτω. Εμείς είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυτού του είδους τα οικονομικά εγκλήματα, ούτως πιν Η ερώτησή μου είναι πιο γενική από αυτή που ήθελα να θέσω που όσον αφορά τη συνεργασία. Έγιναν πολλά βήματα πρόοδου στη διεθνή συνεργασία για να αντιταχθούμε στο οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, τα, εγκλημα τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αλλά και τώρα η κυρία Στεμπόλ είπε ότι δυστυχώ υπάρχει ακόμα πρόβλημα όσον αφορά την ανταλλαγή των πληροφοριών. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, βάσει των εμπειριών σας και τους δύο φιλοξενούμενους μας, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, τι λείπει, τι λείπει ούτω ώστε αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, αυτή η συνεργασία, αυτή η συνεργασία στην οποία πιστεύουμε πολλοί από εμά και εις βάθος μάλιστα, διότι έδωσε άριστα αποτελέσματα. Τι λείπει λοιπόν για αυτή τη συνεργασία. Ε, ένα κοινό φορέα, ε, μια κοινή αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λείπουν οι πόροι, λείπουν νομοθετικέ παρεμβάσει επαρκή. Και εδώ θα το τελευταίο ερώτημα, που είναι πιο γενικό ερώτημα. Έγινε μνήμα και είναι κάτι συγκεκριμένο, το γνωρίζουμε καλά. Ε, αναφέρθηκε, λέγω, πώ αυτέ οι παράνομε συναλλαγέ οικονομικέ χρηματοδότηση τρομοκρατία, αυτέ οι συναλλαγέ βασίζονται στην παράνομη δραστηριότητα των ε, εγκληματιών. Ε, χρησιμοποιούν παραδοσιακέ μεθόδου και πολύ πιο προωθημένε και περίπλοκες. Στην Ευρώπη έχουν εντοπιστεί πάνω από 5.000 οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις και πολλές από αυτές συμμετέχουν στα οικονομικά εγκλήματα και την παράνομη διακίνηση χρήματος και ανακυκλώνουν το χρήμα και αυτό επηρεάζει και την νόμιμη οικονομία των ε, κρατών και γίνεται παράνομο συναγωνισμό των επιχειρήσει κλπ. Θα μπορούσε να έχουμε κοινή έννοια του οργανωμένου εγκλήματο, ένα ορισμό, θα ήταν κάτι χρήσιμο. Δεν υπάρχει και αυτό εμποδίζει και τι έρευνε και τη συνεργασία των κρατών. Θα μπορούσε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση που θα ήταν χρήσιμη με αυτή τη ενία ή τι άλλο. Από την εμπειρία σας λέγω και επαναλαμβάνω. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για να αντικοποιήσουμε αυτή την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών των διαφορών χωρών που είναι το όπλο το ισχυρότερο σίγουρα για να αντιταχθούμε στα εγκλήματα τα οικονομικά και να αντιταχθούμε και στην χρηματοδότηση των ρομοκρατών. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες, ακούσαμε πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο διάλογο. Δεν υπάρχουν ε, άλλοι που θα θέλουν να πάρουν το λόγο, γι' αυτό θα ζητήσω από τον κύριο Ράιζαμπε και την κυρία Ντεμπόλ να απαντήσουν. Έχουν ε, ο καθένας από 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε και να έχουμε τελειώσει στις 11.30 που θα έρθει ο Επίτροπος King, για να συζητήσει μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράισμεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα να πω ότι προσκλήθηκα ως εμπειρογνώμονα της αγγελίας, άρα η δική μου άποψη ενδεχομένως δεν είναι να αντικατοπτρίζει την άποψη της ε, Ολλανδικής κυβέρνησης, είναι κάτι που οφείλω να πω. Άκουσα κάποιες ερωτήσεις που κάνατε σε μένα, απευθύνατε σε μένα. Μιλάτε για την απειλή του κρυπτονομίσματος. Από όσα ε, ασχολούμαι με την ε, καταπολέμηση Τη τρομοκρατία, Πριν από μισό χρόνο ήμουν και πάλι εδώ που έγινε μια συνεδρία σε μια ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία. Ήταν η κυρία Γκόμες παρούσα και ο Ρούσταν Παρόν, ο οποίο έγραψε μια έκθεση για την απειλή του κρυπτονομίσματο για τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, η οποία παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και είχε ζητηθεί και από το Ευρωκοινοβούλιο και το συμπέρασμα αυτής της έκθεσης Ανέφερε αυτά που ήδη είχα πει στην παρουσίασή μου, παρόλο που φυσικά υπάρχει υψηλός κίνδυνος στη χρήση του κρυπτονομίσματος. Στις καθημερινές μας έρευνες δεν το βλέπουμε τόσο όσο θα περιμέναμε να το δούμε. Και εγγυώμαι ότι σε κάθε έρευνα είτε έρευνα σε ηλεκτρονικέ συσκευέ πάντα ψάχνουμε στοιχεία για την ε, χρήση νέων μεθοδών πληρωμών. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, για κάποιο λόγο είτε ψάχνουμε στο λάθος μέρος ή ακόμα βασίζονται περισσότερο στις πιο, πιο παραδοσικές ε, μορφές χρηματοδότησης. Βλέπουμε παραδοσικές μορφέ λοιπόν χρηματοδότηση, ακόμα και αν ε, μας διαφεύγουν οι νέες μέθοδοι πληρωμής βλέπουμε πιο συχνά παραδοσιακέ συναλλαγές. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο, μια άλλη ιστορία όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, όμως αυτό δεν είναι στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για πράγματα που δεν είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο. Είχαμε επιτυχημένες διαδικασίες ενάντια σε απάτες που είχαν να κάνουν με κρυπτονόμισμα. Στην ε, Ολλανδία δεν ε, είναι δύσκολο να γίνει αυτό και γι' αυτό το λόγο μπόρεσαμε να έχουμε επιτυχία στις συγκεκριμένες δίκες. Ένα ερώτημα από την Εστονία αν έχουμε παρομητερική σχέση για το ξέπλυμα του χρηματο όπω και για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας. Το θέμα είναι αν θέλουμε να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα. Στην Ολλανδία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρειαζόμαστε επιγόντως να παρέχουμε τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα μέρη εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την έρευνα και για τη δίωξη. Ένας από τους λόγους που βλέπουμε την έκτακτη αυτή την επίγουσα ανάγκη για την ε, παράδοση των δεδομένων αυτών είναι δύσκολο να αναπτύξουμε αποτελεσματικές τυπολογίες στον εντοπισμό των, ε, των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν ε, τυπολογίες συγκεκριμένε ε, στο, στην παρανομών εσόδων. Υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος για το αν υπάρχει ήδη αυτή η επίγουσα ανάγκη στο να εντοπίσουμε συγκεκριμένες τυπολογίες για τις τακτικές ε, ξεπλήματος χρήματος. Είναι ένας πολιτικός διάλογος περισσότερο αυτός. Οπότε θα περιοριστώ, αλλά για εμάς ε, στις κάτω χώρες είναι ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί υπάρχει ε, το κατεπήγον. Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα απευθύνθηκαν σε μένα. Αν έχω ξεχάσει κάποιο, ευχαριστώ να σα το απαντήσω. Äh, Ευχαριστούμε κύριε Ράιζενμπεκ. Υπάρχουν δύο ακόμα σύντομα ερωτήματα από δύο συναδέλφους. Ο κύριος Μάμαντο από την Πολωνία. Παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με ενδιαφέρει για την απάτη Βίτη και την απάτη καρουσέλ. VPA. Θα ήθελα να ρωτήσω τον διευθυντή της Europol αν έχει γίνει κάτι σε αυτό το τομέα του VAP του ΦΠΑ. Τελική ερώτηση. Από την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Έχετε προβλήματα με τον προπολογισμό για το κυβερνό έγκλημα και την τρομοκρατία, αλλά αν παραμείνει αυτή κατάσταση θα έχουμε μείωση κατά 20 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να απολυθεί προσωπικό, 40 συγκεκριμένα συμβασιούχοι. Πόσα χρειάζεστε πρώτον για να ολοκληρώσετε την αποστολή σας και το δεύτερο όσον αφορά ε, τις αρμοδιότητές σας ε, θα θέλετε να έχετε περισσότερες ή έχει να κάνει με έρευνα, γιατί δεν έχετε ε, ερευνητικές αρμοδιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Ντεμπόλ. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλους για τις σημαντικές σας ερωτήσεις. Θα αρχίσω με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Κοινότητας σε θέματα οικονομικών ερευνών κάθε υπηρεσία επιβολής του νόμου στην Ευρώπη είναι πεπισμένη ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στις έρευνες του οικονομικού εγκλήματος. Αναγνωρίζουν επίσης ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις διάφορες χώρες, ανάμεσα δηλαδή στο επίπεδο των εμπειρογνωμόνων στις διάφορες χώρες ε, μέλη των ειδικών ε, στην νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, στο κυβέρνο έγκλημα κτλ. Οπότε υπάρχουν διαφορές και στην κατάρτιση των ειδικών. Ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν ερευνούμε πάντα οικονομικά όταν υπάρχει σοβαρό έγκλημα. Δηλαδή όταν υπάρχουν σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες ε, δεν σημαίνει ότι πάντα ερευνείται το οικονομικό έγκλημα. Γι' αυτό και είμαστε πεπισμένοι σε επίπεδο Europol ότι χρειάζεται, γιατί μας ρωτήσατε για την ανάκτηση κεφαλαίου, ότι πρέπει να μοιριζόμαστε μεταξύ μας τις βέλτιστες πρακτικές και να τις ανταλλάσσουμε αυτές. Πρέπει να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές λοιπόν και σε αυτό το τομέα και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο γνώσης όσον αφορά την έρευνα του οικονομικού εγκλήματος. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και έχουμε ε, δημιουργήσει μια κεντρική μονάδα στην Europol γιατί έτσι μπορούν να επιβλέψουν καλύτερα όλα όσα συμβαίνουν στο σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό χρειάζεται και το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά τώρα τις παράνομες συναλλαγές στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο, το EC3 που είναι το, η αντίστοιχη μονάδα η ευρωπαϊκή, κάνει έρευνες και προσπαθεί να δει πώς πρέπει να γίνονται οι έρευνες αυτές στο διαδίκτυο και πώς να ανοιχνεύεται η κάθε συναλλαγή. Συνεχίζουμε σε αυτό, αλλά βέβαια πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο η πραγματογνωμοσύνη και να, δίνουμε, και να υπάρχουν συστάσεις που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, τα κέρδη από τη διακίνηση μεταναστών στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα ποσά αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες μας όμως προσπαθούν να ετοιμάσουν μια έκθεση για να υπάρξει μια τέτοια επισκόπηση του τι γίνεται με τα κέρδη από την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τώρα όσον αφορά την πρόταση των κάτω χωρών όσον αφορά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής FIU, θα την εξετάσω την πρόταση. Αλλά όπως ήδη είπα, υπάρχει ένα πρόγραμμα για συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα όσον αφορά τις πληροφορίες ε, σχετικά με το οικονομικό έγκλημα. Είναι ένας ε, πρώτος μηχανισμός που δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Για πρώτη φορά έχουμε κάτι τέτοιο και συμμετέχουν 15 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες και εκπρόσωποι εφαγίου από 8 χώρες. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, είναι ένα πείραμα. Θέλουμε να εκτιμήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εταίρων και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε όσον αφορά την νομική βάση. Να δούμε ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι ώστε να τα αντιμετωπιστούν τα εμπόδια αυτά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό σε αυτό το τομέα είναι εμπιστοσύνη. Γιατί αν έχετε δίκτυα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη οδηγεί στην επιτυχία. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Σε επίπεδο Europol, για παράδειγμα, σκεφτόμαστε έναν κατάλογο ε, στόχων που πρέπει να εμπλέκονται στο θέμα της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία μας στο ΣΟΚ και στο ΣΥΤΙ και είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Όσον αφορά τις απάτες με τα κρυπτονομίσματα και το σύστημα καρουσέλ, έχουμε και εδώ συγκεκριμένα ε, σχέδια. Η Europol παίζει σημαντικό ρόλο. Και όσον αφορά τον προπολογισμό, Πράγματι υπάρχει μείωση. Χτες εξήγησα ήδη τα περί προπολογισμού και σας εξήγησα ποιες είναι οι επιπτώσεις των περικοπών. Οπότε ζητούμε τον ίδιο προπολογισμό όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Η σύσταση της Europol τώρα. Πρέπει να τονίσω ότι πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των πλευρών να υπάρξει δηλαδή μια ευρωπαϊκή, μια πολυμερής εποπτεία. Πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή πολυεθνικό, εν πάση περιπτώσει, επίπεδο. Πρέπει να γίνονται οικονομικές έρευνες και ανάκτηση κεφαλαίων κάθε φορά που έχουμε οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να γίνονται τέτοιες έρευνες δηλαδή. Υπάρχουν σχέδια, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Χτες σας είπα ότι έχουμε τη σύμβαση των επικεφαλής αστυνομιών αυτή τη βδομάδα. Έχουμε συνάντηση επίσης με τις τελωνιακές αρχές και θα το συζητήσουμε. Η ενημέρωση τώρα των μηχανισμών των νομικών δυνατοτήτων που έχουμε για τον εντοπισμό εγκληματικού χρήματος είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει. Έχουμε πληροφορίες, αλλά όχι πάντα τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Και όπως είπε και ο συνάδελφος ε, από τις Ολλανδικές Αρχές, δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε για τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, γιατί πολλέ φορέ πρόκειται για μικρά ποσά, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στι αναφορέ. Άρα πρέπει να ερευνήσουμε περισσότερο και να μπορέσει να υπάρχει ένας πιο ισχυρός συνασπισμός ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στην έρευνα τέτοιων οικονομικών εγκλημάτων. Υπάρχουν πέντε προτεραιότητες για μας τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τις οικονομικές μονάδες, πρέπει να στηρίσουμε τις δράσεις στον πολιτικό κύκλο, ε, και σε αυτό τα λέμε στις χώρες μέλη. Η ανάκτηση κεφαλαιοποίησης πρέπει να ενισχυθεί και αυτό είναι μια δυνατότητα αν συνεργαστούμε περισσότερο με τη Eurojust. Ενισχυμένη επίση συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τέλο πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τι έρευνε που γίνονται για το οικονομικό έγκλημα σε συνεργασία με τι χώρε μέλη. Πρέπει να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να επενδύουμε στη γνώση, στην πραγματογνωμοσύνη, στου ερευνητέ, αλλά και στους ειδικού και στην πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά το διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπόλ και κύριε Ράιζενμπεκ, αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο τέλος αυτού του πάνελ. Σας ευχαριστώ που πήρατε το λόγο και θέσετε αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντικό να οικοδομήσουμε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη προς την κυρία Ντεμπόλ για να καταπολεμήσουμε τις διαφορετικούς τύπους εγκλήματος. Ο κύριος Κίνγκ θα είναι μαζί μας στις 11.30, άρα να σας ζητήσω να μείνετε στην αίθουσα για να ξεκινήσουμε με το επόμενο πάνελ στις 11.30. Ευχαριστώ πολύ. Would Πρόεδρε, μου επιτρέπετε μία ερώτηση να κάνω στην κυρία Ντεμπόλ, μια που έχουμε χρόνο. Μπορείτε, αλλά ιδιαίτερος. Μα μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα η ερώτησή μου όλους. Μα τελειώσαμε την, ε, το κομμάτι αυτό της συνάντησης. So we

Yeah, I, I...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 Dear colleagues, let's start our next panel. Πάμε λοιπόν στο επόμενο πάνελ. Ich freue mich sehr. Χαίρομαι πολύ που μας κάνει την τιμή ο Επίτροπος Κίνγκ στην ε, μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα μας μιλήσει για την τρέχουσα κατάσταση και τις ε, προόδους που έχουν σημειωθεί για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον ρόλο επίσης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Επίτροπε Κίνγκ, θα μάθουμε λοιπόν από εσά τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα ασφαλείας. Ο λόγο σε εσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που επέστρεψα σε μία από αυτές τις συνεδριάσεις. Χαίρομαι. Χαίρομαι που διεξάγονται και οργανώνεται αυτές τις συναντήσεις. Αυτού του είδους ο συλλογικός έλεγχος και συμμετοχή και διάλογος είναι σημαντικός. Όχι μόνο για την Ευρωπόλ, αλλά για όλους μας που συμμετέχουμε σε αυτές τις εργασίες, σε συνεργασία με την Europol, για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά προβλήματα, τα σχέδια για να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα μελλοντικά προβλήματα. Η συμμετοχή σας βοηθά εμάς να σχεδιάζουμε καλύτερα και κατάλληλα τα μέτρα και να στηρίζουμε την Europol στις προσπάθειες που καταβάλει στον τομέα αυτόν. Ελπίζω ότι θα δεχτείτε ότι δεν χρειάζεται να πιστώ εγώ για το πόσο σημαντική είναι η Europol. Εγώ είμαι ένθερμος υποστηριχτής στη Europol. Πιστεύω ότι είναι σημαντικός φορέας. Πιστεύω στο έργο της Europol. Χρειάζομαι ότι θα πρέπει να δώσουμε σωστή στήριξη στο έργο αυτό. Οικονομική στήριξη αλλά και μέσω πολιτικών και μέσω εργαλείων. Είναι σημαντικό το ότι συζητήσαμε κάποια από τα εργαλεία πολιτικής που μπορούμε να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε για να βοηθήσουμε την Europol να πετύχει το στόχο της προς το συλλογικό καλό, δηλαδή την ασφάλεια όλων μας. Με καλέσατε νομίζω να σας ενημερώσω συντομία για τις εργασίες που έχουμε κάνει πρόσφατα όσον αφορά τα θέματα της ε, Ένωσης Ασφαλείας μετά από αυτά που είπαμε στη συνεδρίασή μας επί Βουλγαρικής Προεδρίας στην Άνοιξη, συνεχίσαμε τις εργασίες μας στο θέμα αντιμετωπίσης τρομοκρατίας, στα προβλήματα στον κυβερνοχώρο, κυβερνοαπειλές και απειλές που θα χρησιμοποιήσουν τον κυβερνοχώρο και σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, υβριδικές απειλές συζητήσαμε και απειλές από χημικά, βιολογικά, πυρηνικά, ραδιολογικά, ραδιολογικές πηγές, κάτι που δεν είναι ένα αφηρημένο θεωρητικό πρόβλημα. Το είδαμε αυτό στο Σόλσμπερι, στη χώρα μου. Τι συνέβη στο Σόλσμπερι. Και πρόσφατα ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε αρκετές νέες πρωτοβουλίες σχετικές με την Ένωση Ασφαλείας στη δική του ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τα είπε αυτά αρχές του μηνός Ξεκινώ λοιπόν από εκεί, τις προτάσεις αυτές. Μεταξύ αυτών των προτάσεων υπήρχε και μία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. απευθυνόμενη προς τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο για την καταπολέμηση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυτό το πρόβλημα των τρομοκρατικών προκλήσεων στο διαδίκτυο είναι πραγματικό κίνδυνο ε, όσον αφορά την ασφαλειά μας. Τον Ιανουάριο του 2018 και μόνο περίπου 700, 700 νέες τέτοιες αναρτήσεις προπαγάνδα του ISIS ή DICE είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Το τρομοκρατικό περιεχόμενο ενετοπίστη από τη Europol, που είναι το κέντρο αριστείας και γνώσεως σε αυτό το τομέα, σε πάνω από 150 πλατφόρμες αυτός είναι ένας ε, πραγματικός κίνδυνος προς αντιμετώπιση. Λοιπόν, το περιεχόμενο το νομοκρατικό στο διαδίκτυο έπαιξε ρόλο σε κάθε μία από τις επιθέσεις που έγιναν στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Είτε μέσω παρακίνησης να διαπραχθούν οι επιθέσεις, είτε μέσω οδηγιών σε κάποιες περιπτώσεις σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, είτε συχνά μέσω ε, τρομοκρατικής επιθέσεως και των φρικτών αποτελεσμάτων. Συνεργαστήκαμε με τις μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου επιθελοντικής βάσεως ε, για κάποια χρόνια. Συμμετείχαν και εκπρόσωποι των κρατών μελών και εκπρόσωποι της Europol και αυτό ήταν σημαντικό στο, στο φόρουμ για το διαδίκτυο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Λοιπόν, η Europol εντόπισε περίπου 6.000 ε, περιπτώσεις τρομοκρατικού περιεχομένου σε πάνω από 130 ε, διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών και έδωσε αναλυτική και επιχειρησιακή υποστήριξη στα κράτη-μέλη, τις αρχές των κρατών μελών, κυρίως μετά από κάποιες από τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις και αυτές οι προσπάθειες, οι λογικές προσπάθειες, εδραζόμενες επί της τεχνογνωσίας της Ευρωπόλ έδωσαν θετικά αποτελέσματα. Αλλά η πρόοδος πεπετεύχθη εντός του φόρουμ εθελοντικός δεν πήγε αρκετά μακριά, δεν προχωρήσαμε αρκετά μακριά, αρκετά γρήγορα. Υπάρχει πάρα πολύ περιεχόμενο ακόμα εκεί, στο διαδίκτυο. Κάναμε ένα βήμα λοιπόν, για πρώτη φορά, και προτείναμε νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δημιουργεί υποχρεώσεις που θα υπέχουν όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και άμεσα και οι πλατφόρμες για αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος, αυτής της απειλής. Οι προτάσεις μας που απεκάλυψε ο κύριος Γιούνκερ, ο πρόεδρος Γιούνκερ, θα δημιουργήσουν τρεις υποχρεώσεις, νέες υποχρεώσεις. Υποχρέωση που υπέχει η πλατφόρμα θα είναι υποχρεωτικό οι πλατφόρμες να κατεβάζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο εντός μιας ώρας μετά την παραλαβή συγκεκριμένης εντολής αφαίρεσης από την αστυνομία ή τις δικαστικές αρχές. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι όπως γνωρίζουμε το τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι άκρος επιβλαβές τις πρώτες ώρες μετά την εμφάνιση στο διαδίκτυο, διότι διαδίδεται και έρευνα που κάναμε κατέδειξε τα τρία τέταρτα όλων των διασυνδέσμων με την προπαγάνδα του ΝΤΕΣ ε, μοιράζονται μέσα σε τρει ώρε από την ανάρτηση. Αν κόψουμε πολύ νωρίτερα αυτό το κύκλο, ε, είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα. Δεύτερον, αν μια πλατφόρμα έχει αποδειχτεί, είναι προφανές, ότι χρησιμοποιείται για διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ενεργά μέτρα προς εντοπισμό του περιεχομένου και πρόληψη ε, επανανάρτησης ή ανάρτησης αυτού και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέσουν επαρκείς πόρους ούτως ώστε αποτελεσματικά να εντοπίζουν τρομοκρατικό περιεχόμενο και να εκδίδουν εντάλματα ε, αφαιρέσεως του περιεχομένου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε βεβαίως ότι υπάρχουν και μέτρα διαφύλαξης ισχυρά όπως δυνατότητες υποβολής καταγγελιών και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής αν αυτό παραστεί αναγκαίο διότι Αυτές οι προτάσεις δεν αφορούν λογοκρισία. Θέλουμε να στοχεύσουμε παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο, περιεχόμενο που θα ήταν παράνομο και εκτός διαδικτύου και επί του διαδικτύου. Η τεράστια πλειοψηφία των πλατφορμών συνεργάζεται και θα συνεργαστεί, αλλά χρειαζόμαστε διατάξεις για αποτελεσματικές κυρώσεις και γι' αυτό προτείνουμε τη δυνατότητα σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης με εντάλματα αφαίρεσης όχι μόνο πρόβλημα σε μια περίπτωση, με άλλα λόγια δύο περιπτώσεις, αλλά συστηματική μη συμμόρφωση σε περίπτωση τέτοια να έχουμε σημαντικές κυρώσεις που θα μπορούν να επιβληθούν σε πάροχο υπηρεσιών μέχρι 4% ε, του παγκόσμιου κύκλου εργασιών, όπως προβλέπεται και από το GDPR σε κυρώσεις. Και αυτό σε συνεχή συνεργασία που υπάρχει ε, με όλους τους εμπλεκομένους φορείς αν συνεχιστεί αυτό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κρίσιμο πρόβλημα αυτό που είναι ένα εργαλείο στο πλωστάσιο των τρομοκρατών. Δεν μιλάμε για λογοκρισία, δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη, αλλά για υλικό που παρακινεί ή προωθεί τρομοκρατικές πράξεις ή εξυμνεί τρομοκρατικές ομάδες ή δίνει οδηγίες για την παραγματοποίηση επιθέσεων. Αυτό είναι παράνομο και στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου είναι περιεχόμενο πρέπει να αφαιρεθεί όπου και να βρίσκεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τμήμα του φάσματος των απειλών που αντιμετωπίζουμε στον κυβερνοχώρο και γι' αυτό όμως, επειδή έχουμε βρει φάσμα απειλών, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για να εξασφαλίσουμε καλύτερο τρόπο την ασφάλεια των εκλογών μα και των δημοκρατικών μα διαδικασιών. Οι προτάσει δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουμε και να δυναμώσουμε την ασφάλεια των εκλογικών διαδικασιών, διότι επίκυνται διάφορες εκλογές σε διάφορα κράτη-μέλη τους επόμενου μήνες και βέβαια εν ώψη των επικειμένων ευρωεκλογών τον επόμενο Μάιο. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους και να έχουμε ετοιμαστεί. Αυτά περιέχουν συστάσεις για καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, για να υπάρχει συνεργασία, δίκτυο, συμμετοχή αρμόδιων αρχών, φορείς προστασίας των δεδομένων και να δημιουργήσουμε ε, ένα δίκτυο συνεργασίας για τις εκλογές. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και θέλουμε οι εθνικές αρχές και τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα να λάβουν μέτρα να προστατεύσουν τα δίκτυά τους από παρεμβάσεις στο διαδίκτυο. Και είχαμε κάνει και άλλες εργασίες για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο εστιαζόμενη τη αυτή περιπτώση προσπαθειών παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ζητήσαμε τις πλατφόρμες να δραστηριοποιηθούν για βελτίωση ανεχνεσιμότητα, λογοδοσία και διαφάνεια στο διαδίκτυο και να προστατευτούν καλύτερα οι χρήστε. Περιμένουμε μαζί με τι πλατφόρμες τι επόμενε ημέρε να δημιουργήσουμε δεδολογικό κώδικα για αυτά τα θέματα. Μπορεί να γίνει διαφορά. Στη, στη μάχη πρέπει να κερδίσουμε. Διαφορετικά, αυτοί που θέλουν να παρέμβουν στι δημοκρατικέ διαδικασίε μα θα ρίξουν σκιά σε αυτές και θα υπονομεύσουν την αξιοπιστία που θέλουμε να έχουν οι διαδικασίες. Χρειαζόμαστε όλοι οι φορείς να συνεργαστούν στενότερα και προτείνουμε να δημιουργηθούν αυτά τα δίκτυα συνεργασίας. Αυτό θα βοηθήσει. Και ελπίζω, σαν αυτού, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε βασιζόμενοι επί του κέντρου εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας του Europol για να αντιμετωπίσουμε διάφορες πτυχές των κυβερνών προβλημάτων επόμενο βήμα διάσκεψη ψηλού επίπεδου της Task Force για την Ασφάλεια εδώ στις Βρυξέλλες 15-16 Οκτωβρίου συζητήσουμε συγκεκριμένους τρόπους για καλύτερη αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, απειλών ενώπιον των εκλογών για τις κυβέρνο Εδώ και ένα χρόνο δώσαμε ένα πακέτο προτάσεων για την ενίσχυση της κυβέρνων βάσει τριών πυλώνων αντοχής, αποτροπής και διεθνούς συνεργασίας και άμυνας. Σημειώσαμε έκτοτε καλή πρόοδο επ' αυτό. Να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη για μεγαλύτερη εντοχή. Θα είμαστε πιο δύσκολο να δεχτούμε επίθεση και να τα ταχύτερα, δημιουργώντας πραγματική υπηρεσία κυβερνοασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θεσπίσει πρότυπα και να ανταποκρίνεται σε επιθέσεις κλίμακας, εδραζόμενη επί της εμπειρίας της ΕΝΙΣΑ. Ο φορέας αυτός θα αντιμετωπίζει θα έχει χρέη ανταπόκριση κρίση, να αντιμετωπίσει κυβερνοεπιθέσει και να δημιουργήσει σχέδιο συνεργασία για τη μετώπιση τέτοιων επιθέσεων με συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Έτσι θα ενισχύσουμε τη συλλογική απάντηση σε επιθέσει κλίμακα στον κυβερνοχώρο και θα έχουμε σωστό σχέδιο δράση προγραμματισμένο. Πρέπει να συνεργαστούμε αρχέ κρατών μελών και υπηρεσία κυβερνοασφαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι το σχέδιο που θα καταρτήσουμε θα είναι λειτουργικό, επιχειρησιακό και δοκιμασμένο. Μετά από διάφορες ασκήσεις, η υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για πρότυπα και επιστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κυβερνοασφάλεια και τα προϊόντα και υπηρεσίε θα πληρούν τα στα επίπεδα ασφαλεία. Στόχο τη προσεγγίσεω για την πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεργαστούμε με τις αρχές των κρατών μελών και θα τα κοπρινόμεθα σε διάφορες ανάγκες ασφαλείας, σε διάφορους τομείς. Πιστεύω ότι στον αένα διασυνδεούμενο κόσμο χρειαζόμαστε ευέλικτο πλαίσιο πιστοποίησης όχι μόνο για να δημιουργήσουμε ψηλά πρότυπα και μόνο, να δημιουργήσουμε έναν θετικό κύκλο, ούτω ώστε η κυβερνοασφάλεια να έχει ύψιστη προτεραιότητα για τον ιδιωτικό τομέα, τι επιχειρήσει, καθώ και το δημόσιο τομέα και του φορεί αυτού και να είναι πηγή δημιουργία εμπιστοσύνη και με εμπιστοσύνη και να έχουμε και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα είναι κρισίμου σημασία να κάνουμε τα αναγκαία βήματα για να βελτιώσουμε την αποτροπή στα πλαίσια της κυβερνοασφάλειας και εδώ βασικό ρόλο παίζει η Europol και το EC3. Πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματικά αντικίνητρα, πιστικά αντικίνητρα για αυτούς που θέλουν να μας επιτεθούν. Πρέπει δραματικά να αυξήσουμε τις πιθανότητες να πιαστούν αυτοί και να λογοδοτήσουν. Με αυστηρές κυρώσεις που θα επιβληθούν σε εκείνους που θα επιτίθενται μέσω του κυβερνοχώρου. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κρίσιμο ρόλο να παίξουν για να ειχνεύσουμε να εντοπίσουμε τους ε, ε, αυτούς που διαπράττουν αντικείμενα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όπως γνωρίζετε από την πόλη 90% των κυβερνοεγκλημάτων πολύ συχνά δεν εξηχνιάζονται. Υπάρχουν προβλήματα. Having a transparent way of tracing websites and Υπάρχουν βασικοί τομεί όπω είναι οι, ικανότητε να εντοπίζουμε το κυβερνό έγκλημα. Είναι θέμα σημαντικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από το κυβερνό έγκλημα είναι πολύ βασικό για το μέτωπο πληροφοριών και για την υποστήριξη των κρατών μελών και των αρχών τους ε, για τις έρευνες, ε, την επιχειρησιακή ανάλυση, τον συντονισμό και την εμπειρογνωμοσύνη. Και έχει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία που είναι αναγνωρισμένη από όλα τα κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Παραδείγματο χάρη την άνοιξη φέτος, η μεγαλύτερη αγορά που δέχτηκε επιθέσεις και που χάρη στη συνεργασία δίντος επιθέσεις κατάφερε ε, να το αντιμετωπίσει με τη βοήθεια της Europol. Το κόστος των επιθέσεων αξιολογήθηκε στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια μικρή συνασφορά αν αναλογιστούμε το μέγεθος της πρόκλησης αυτής που συνεχίζει να υπάρχει στο κυβερνό έγκλημα και κάναμε βήματα του ώστε οι δυνάμει του νόμου να μπορεί συλλέγει πιο εύκολα τα στοιχεία για να λογοδοτήσουν οι εγκληματίε, ηλεκτρονικά στοιχεία που πολύ συχνά βρίσκονται στοιχεία σε διαφορετική δικαιοδοσία. Αρχέ του έτου δημιουργήσαμε προτάσει ούτω ώστε οι δικαστικέ αρχέ και οι δυνάμει του νόμου να έχουν νέα εργαλεία που χρειάζονται ούτω ώστε να αποκτήσουν στοιχεία διασυνοριακά, ε, email, κείμενα, μηνύματα WhatsApp, ηλεκτρονικά μηνύματα για έρευνα και για δίωξη εκείνων που διαπράττουν εγκλήμα, τρομοκρατία και άλλα σοβαρά εγκλήματα του οργανωμένου εγκλήματος ταχύτερα, πολύ ταχύτερα από ό,τι μπορούν να κάνουν τώρα. Αυτή τη στιγμή, με συστάμενους κανόνες και διαδικασίες, μπορεί να χρειαστούν οι δυνάμει του νόμου περίπου κατά μέσο όρο 10 μήνε για να αποκτήσουν αυτά τα στοιχεία όταν βρίσκονται τα στοιχεία αυτά σε μια άλλη δικαιοδοσία και οι προτάσεις μας έχουν σχεδιαστεί ούτω ώστε ριζικά να μειώσουν και να αλλάξουν αυτή την προσπάθεια ώστε αυτά τα στοιχεία να μπορούν να αποκτηθούν σε δεκαήμερο ή και έξι ώρες σε περίπτωση επιγόντων περιστατικών. Κάποια λόγια τώρα για την καταπολέμηση της χρηματοδοτήσεως των δρομοκρατών και το ξέπλυμα χρήματος. Εφόσον τα συζητήσατε αυτά τα θέματα, και ήταν ένα από τα βασικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει περαιτέρω ενίσχυση τη εποπτεία των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων τη Ευρωπαϊκή Ενώση για να αντιμετωπιστεί καλύτερα το θέμα του ξεπλήματο χρήματο και των απειλών ε, των τρομοκρατικών εν γέννη, ενισχύοντα ε, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να έχει τα αναγκαία εργαλεία και πόρου για να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία και σύγκληση εποπτικών προδιαγραφών στον ε, τομέα που εποπτεύει. Ένα τμήμα ευρύτερη στρατηγική να ενισχυθεί το πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ενώσεω για προληπτική εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματο από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Έτσι θα προωθήσουμε την ακαιρεότητα του χρηματοστικού συστήματο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα εξασφαλίσουμε χρηματοστική σταθερότητα και θα αυξηθεί η προστασία μα από το οικονομικό έγκλημα. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε να εστιαζούμε τις προσπάθειες κατά συγκεκριμένου προβλήματος της χρηματοδοτήσεως των τρομοκρατών. Μια εποχή που μιλάνε κάποιοι για τρομοκρατία low cost και μοναδικούς, μοναχικούς λύκους που επιτίθενται, θα ήταν εσφαλμένο να εγκαταλείψουμε την χρήση της συλλογή οικονομικών στοιχείων κατά της τρομοκρατίας. Παραμένει πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο Κάναμε προτάσει αρχέ του έτου, ούτω ώστε οι δυνάμει του νόμου να μπορούν έγκαιρα έχουν πρόσβαση σε οικονομικέ πληροφορίε που είναι απαραίτητε για την εξυχνίαση διάφορων σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης τη τρομοκρατία, πληροφορίε για τραπεζικού λογαριασμού και να γίνεται και οικονομική ανάλυση και τα στοιχεία αυτά να μπορούν να τα έχουν διαθέσει του. και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ εθνικών φορέων και εθνικών μονάδων συλλογή οικονομικών στοιχείων και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών πρέπει να λαμβάνει η χώρα με την υποστήριξη για δημιουργία ενός δικτύου ε, μονάδων συλλογής οικονομικών στοιχείων. Και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν διαδικασίες επ' αυτών γρήγορα, διότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Κάνοντας αυτό, πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά, το επόμενο βήμα. Κατά την άποψή μου, πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο πρέπει να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Σύστημα ανίχτευση Χρηματοδότηση Τρομοκρατών. Κάτι που θα συμπληρώνει την έξω συνεργασία που απολαμβάνει η Europol με του Αμερικανού εταίρου και το δικό τους πρόγραμμα για την ε, ταυτοποίηση και εντοπισμό τρομοκρατικών ε, δρόμων χρηματοδότησης. Καμιά φορά ο καλύτερος τρόπος για να μαζέψουμε αυτά τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση για τους Ευρωπαίους πολίτες, αν και είναι παράδοξο, είναι να περάσουμε μέσω των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς νομίζω ότι αυτό είναι παράδοξο. Πρέπει να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι να το κάνουμε μόνοι μας, βασιζόμενοι επί της εμπειρίας της ε, Europol. Όσον αφορά την ασφάλεια, θα πρέπει να δούμε και πέρα από τα σύνορα αστάθεια στην περιοχή μας μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τη δική μας εσωτερική μας ασφάλεια, το ξέρουμε αυτό και γι' αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χώρες στη γειτονιά μας ούτως ώστε να αυξήσουν τις δυνατότητες πονεμής τρομοκρατίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος με βασικό ρόλο να παίξουν οι διάφοροι φορείς μας, το Eurojust, η Σεπόλ και άλλοι και κυρίως η Europol Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να ευχαριστήσω τη Europol μέσω της ηγεσία αυτής για το έξοχο έργο της Europol που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις δυνάμεις, τους φορείς των κρατών μελών και άλλους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια και αλλού ε, στη γειτονιά μας σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι από κοινού πολεμάμε το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος κυρίως το παράνομο εμπόριο πυροβόλων όπλων και άλλες πτυχές ε, που αφορούν τη συνεργασία για την ασφάλεια διατηρώντα ισχυρή συνεργασία με τέρου όπω η ΕΠΑ ταυτόχρονα και τον Καναδά. Βελτιώνουμε τη συνεργασία μα με διεθνεί φορεί για διάφορα θέματα όπως αντιμετώπιση ε, και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Τέλο του προηγούμενου έτου παρουσιάσαμε συστάσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσει για διεθνεί συμφωνίε μεταξύ Ευρωπόλ και διαφόρων χωρών εταίρων επιτρέποντας ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων με αυτές τις χώρες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε σταθερή ε, πρόοδο στις συνεργασίες μας, για τη συνεργασία μας, διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται η διαπραγματεύση αυτών των συμφωνιών. Είναι θέμα επιχειρησιακό, επιχειρησιακή ανάγκη. η συνεργασία των ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων είναι κάτι που χρειάζεται ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των ξένων μαχητών, των δρομοκατών αυτών, και κάποιου υπόπτου που μπορεί να έχουν διπλή υπηκότητα η νόμιμη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε τρίτες χώρες. Χρειάζεται στενότητα συνεργασία αρχών του νόμου για να εντοπίσουμε και να διώξουμε τρομοκράτε και εγκληματίες και να εντοπίσουμε και να αποφύγουμε το ταξίδι τρομοκρατών, την κατάχρηση του διαδικτύου από του τρομοκράτε και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Αυτέ οι διεθνεί συμφωνίε έχουν πρόθεση να θεσπίσουν μέτρα διαφύλαξης όσον αφορά την προφύλαξη των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων για να διευκολύνουμε την επιχειρησιακή συνεργασία. Και τα στηρίζουμε. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ό,τι πρόοδο επιτευχθεί σε διαπραγματεύσεις. Και πολύ χαίρομαι σε επόμενες συναντήσεις του σώματος αυτού να σας ενημερώσω. Και για να ολοκληρώσω, Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Europol για το εξαίρετο έργο τους το τελευταίο διάστημα. Καθημερινά προωθούν τις προτεραιότητες και στηρίζουν τις χώρες μέλη και τις ε, εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και φροντίζουν και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ε, του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. King, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε Κίνγκ για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Ο κύριος Διαθ τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ως ήθιστε, πάντα έχετε να μας πείτε κάτι σημαντικό όσον αφορά την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Τώρα κάποια πράγματα για να κλείσουμε μετά την παρουσίασή σας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που τονίζετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Europol. Εδώ έχουμε το άρθρο 88 και το άρθρο 51 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούν για τον κοινοβουλευτικό αυτό έλεγχο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή στην Europol για αυτήν την τόσο σημαντική υπηρεσία που είναι η Europol. Πράγματι, η Europol, ε, κύριε Πίτροπε, χρειάζεται μηχανισμούς, χρειάζεται βοήθεια έτσι ώστε να υλοποιήσει την Ένωση της Ασφάλειας που είναι αυτή η υπέροχη ιδέα της. Και γι' αυτό όμως χρειάζεται πρικοδότηση, χρειάζεται μέσα. Απαιτούμε πολλά. Η τρομοκρατία ε, επιγραμμικά, online. Ξέρουμε ε, το περιεχόμενο πόσο γρήγορα κυκλοφορεί από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. Είναι γνωστό Χρειαζόμαστε λοιπόν μέσα, προσωπικό, κατάρτιση και χρήματα. Η δήλωση του Προέδρου Γιούνκερ να σβήνονται κάποια περιεχόμενα μέσα σε μία ώρα είναι κάτι εφικτό, αλλά χρειάζεται μέσα, προσωπικό και χρήματα. Μια εξαιρετική ιδέα επίσης που έχει να κάνει και με τις εκλογές όπου μερικές φορές η κυκλοφορία περιεχομένου πλήττει την ε, ανεξαρτησία. Συνεπώς πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα μέσα που διαθέτουμε, το EC3 για παράδειγμα, και η ασφάλεια, μην ξεχνάμε ότι έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Οι κακοί πρέπει να μας φοβούνται εξαιτίας των μέσων που διαθέτουμε. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές διασυνοριακά πρέπει να εντοπίζονται γρήγορα εφόσον είναι ύποπτες. Εσείς το είπατε πολύ σωστά. Κύριε Επίτροπε, Πράγματι, αφιερώσαμε χρόνο και συζήτηση σε θέματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και πράγματι μας απασχόλησε και μας πόνεσε η διαπίστωση ότι μερικές φορές η τρομοκρατία μπορεί να υπάρχει και χωρίς κόστος και να χτυπάει όμως και να προκαλεί τόσο πόνο. Συνεπώς, οι ε, μυστικές πληροφορίες, υπηρεσίες πληροφοριών όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές πρέπει να λειτουργεί καλά. Έχουμε το ευτυπιστή οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο και στην Ευρώπη. Τέλος, οι διεθνείς συμφωνίες είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος γενικά. Αλλά βέβαια τέτοιες συμφωνίες πρέπει πάντα να τηρούν όσα ισχύουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για τόσα μας είπατε. Τώρα πρέπει να σας κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σαν συμπεράσματα, όχι, δεν προβλέπετε παρεμβάσει μετά την παρουσίαση του Επιτρόπου. Είμαστε στα συμπεράσματα. Λοιπόν, όσον αφορά τα συμπεράσματα για τις εργασίες μας, χθες και σήμερα, πρέπει να σας πω ότι θα διατυπωθούν με ακρίβεια και θα ανακοινωθούν στην επόμενη συνάντηση στο, στο Βουκουρέστι. Τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνουν τέσσερα σημεία. Το ένα έχει να κάνει με το πρόγραμμα εργασίας της Europol. Το πρόγραμμα αυτό εργασιών της Europol συνδέεται επιμένω με την κατάλληλη πρικοδότηση ε, στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεύτερον, προστασία δεδομένων. Και αυτό θα διατυπώνεται συγκεκριμένα στα συμπεράσματά μας. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε εκτενώς για αυτό το ζήτημα. Και τέλος, συνεισφορά της Europol στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, στην ανάκτηση κεφαλαίων και την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Και βέβαια τόσα μας είπε ο Επίτροπος Κίνγκ. Επιπλέον θέλω να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στο Βουκουρέστι 24 και 25 Η ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου επίσης θα συνεχίσει τις εργασίες της μέχρι το Φεβρουάριο του 2019. Θέλω επίσης να ενημερώσω για την ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε προκειμένου η Δανέζικη αντιπροσωπεία να μπορέσει να προσφέρει συγκεκριμένες συστάσεις για τους ε, κανόνες διαδικασίας στην νέα αυτή ομάδα. Είχαμε μια διμερή συνάντηση με τη δανέζικη αντιπροσωπεία που ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα και μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Η Δανία, όπως πάντα, πρέπει και τώρα να παίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των Ευρωπαίων. Με αυτά λοιπόν, Πρόεδρε, εφόσον μου επιτρέπετε, θα σας ζητήσω να Κυρίσετε εσεί τη λήξη τη συνεδρίασης αυτής. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι, σα έχουμε φτάσει στο τέλος της συνεδρίασής μας. Με πολύ ωραίο τρόπο συζητήσαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συζητητές και από χθε και ιδιαίτερα τον Επίτροπο για την ε, παρουσία του ο Σάρφος Διά Δεμέρα έχει αναφερθεί ήδη στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει τον Φεβρουάριο στο Βουκουρέστι. Ελπίζω και εκεί να έχουμε έναν εξίσου ενδιαφέρον διάλογο και να ε, δούμε και τι συμβαίνει από πλευρά δανέζικης αντιπροσωπείας. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην συνεδρίαση αυτή την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, τις ε, υπεύθυνε αρχές, τα Εθνικά Κοινοβούλια, τους Ιερμηνείς και τους ε, συνεργάτες της ε, Αυστριακής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και σας εύχομαι καλή παραμονή στις Βρυξέλλες και ασφαλή επιστροφή στι πατρίδα σας. Ευχαριστώ πολύ. To Μία ανακοίνωση για το Βουκουρέστι θέλω να κάνω παρακαλώ. Συγγνώμη, εδώ. Θέλω να κάνω μία ανακοίνωση σε σχέση με τη συνάντηση στο Βουκουρέστι. Ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Να ξέρετε ότι σήμερα το πρωί το Ρουμανικό Κοινοβούλιο στο Βουκουρέστι για να μεταφέρει τη, στην Εθνική Νομοθεσία το άρθρο 4 για την ε, νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος ε, αφαίρεσε το κομμάτι για το ΠΕΠΣ. Οπότε, εν ώψη της συνάντησης αυτής στο Βουκουρέστι, ίσως θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας κατά πόσο δηλαδή στη Ρουμανία Όντω γίνεται προσπάθεια για την καταπολέμηση της νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Μήπω η ρουμανική αντιπροσωπεία θέλει να απαντήσει σε αυτό κάτι, πέντε δευτερόλεπτα έχετε. Όχι.